Euh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, euh, euh, συνεχίζουμε τις εργασίες του εργαστηρίου μελέτη μας με θέμα την ελεύθερη διακίνηση των ε, πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που λαμβάνουν μέρος ε, στο σεμινάριο. θα δώσω το λόγο στον Κιούρτ Λέχνερ και την Αλεξάνδρα Θέιν για τις εναρκτήριες ομιλίες τους ε, στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου που έχει τίτλο «Οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο». Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Κούρτ Λέχνερ, που είναι πρώην μέλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Τον ακούμε κύριε Λέχνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ και πάλι μεταξύ σας, διότι έχω έξι μήνες να έρθω στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι μετά από δύο, τρία χρόνια ε, ενασχόλης ως ε, εισηγητής είχα εξαντληθεί και έπρεπε να ξεκουραστώ. Ήταν πολύ κουραστικό, αλλά νομίζω πολύ ε, επικοδομητική αυτή μου η ε, προσπάθεια και είχε καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι άξιζαν ε, οι συζητήσεις που κάναμε. Παραλαμβάνω την πρόταση της Επιτροπής. Παραλαμβάνω ότι ήταν καλή πρόταση της Επιτροπής. Αλλά ε, μέσω των συζητήσεων βελτιώθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη και αυτό θέλω να πω και τα τρία θεσμικά όργανα συμμετείχαν σε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι έχουν γίνει έκτοτε διάφορες συνδιοργανώσεις, έχουν τεθεί ερωτήματα, όπου και εγώ, και εγώ συμμετείχα. Γιατί είναι τόσα τα προβλήματα που έχουν προκύψει, για να μην θεωρηθείτε είμαι υπεύθυνο που δεν τα επίλυσα, επέλυσα με τις προσπάθειες που είχα κάνει. Έχουμε πολλά προβλήματα. Η ελεύθερη διακίνηση, και ένα σωστό κληρονομικό δίκαιο και να αναφερθώ σε κάτι πολύ απλό στο Βέλιο και στη Γαλλία για τα ακίνητα υπήρχε πάντα το lex resite δηλαδή το, τα γαλλικά θέματα ακινήτων ε, ε, ρυθμίζονται με βάση το γαλλικό δίκαιο, οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα. Και το εμπράγματο και το δίκαιο για την καταχώρηση έχουν ε, ε, συντονιστεί μέσω προσπάθειας ναι, προσπάθειες εναρμόνισης, αλλά τώρα, λόγω νέων καταστάσεων, έχουν προκύψει νέα προβλήματα. Γι' αυτό σήμερα το πρωί όταν συζητάγαμε για το εμπράγματο θεωρώ ότι πρέπει να συντονιστούν ορισμένα αλλά δεν είναι δυνατόν να είμαστε υπερβολικοί, δεν είναι δυνατόν όλα τα ε, δίκαια να συντονιστούν. Πιστεύω όμως ότι τα θέματα που σχετίζονται με, τη, με τις κληρονομίες μπορούν να συντονιστούν. Όπου ε, συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις, ε, ε, βλέπω ότι ο κανονισμός αυτός ε, δεν αντιμετωπίζεται πολύ θετικά και αρνητικά σχόλια δεν έχω ακούσει, μόνο κάποια συγκεκριμένα σχόλια. Προς την Κομισιόν θέλω να πω, να κάνω την παράκληση, να προσπαθήσουν ότι όταν θα εκπονήσουν τα διάφορα έγγραφα να προσπαθήσουν, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτω ώστε να είναι αρκετά σαφή. Δεν είναι να το αναβασιστούμε σε εθνικές διαδικασίες. Μην επιτρέψετε οποιοδήποτε έτοιμα κράτους μέλους να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί στα έντυπά σας, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να είναι τόσο περίπλοκο το έντυπο που θα προκύψει που να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν πλέον καλά. Χρειαζόμαστε βεβαίως αποφάσεις. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει νομική σαφήνεια. Υπάρχουν πολλά ε, επιμέρους προβλήματα που ήταν αναπόφευκτα. Ορισμένα θα μπορούσαμε όμως να τα έχουμε αποφύγουμε αλλά πολλές φορές ε, οι σύγχρονοι νομοθέτες θέλουν να, να ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες. Δεν είναι δυνατόν ε, μέσω ενός νομοθετήματος να τα ρυθμίσουμε όλα. Χαίρομαι που θα μας μιλήσει και ο καθηγητής ε, Χες μετά και ελπίζω ότι δεν πήρα πολύ από το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε αγαπητέ Κουρτ για την παρουσίαση. Τη σκητάλη στη νομική επιτροπή για το θέμα που ήσουν αρμόδιος εσύ την έλαβε η Αλεξάνδρα Τέιν. Της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι εάν οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας διακίνησης. Και πρέπει να πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η απάντηση είναι όχι, αν και είναι λυπηρό. Είμαι εισηγήτρια για, τις δύο, για τους δύο κανονισμούς για τα περιουσιακά στοιχεία. Ε, ο ένας κανονισμός αφορά ε, τους γάμους που μπορεί να είναι και μεταξύ ομοφύλων ε, καθώς και τις, συγγνώμη, τις καταχωρημένες εταιρικές σχέσεις που μπορεί να είναι μεταξύ ομοφύλων και τους γάμους. Για το θέμα αυτών των ομοφύλων καταχωρημένων σχέσεων βλέπουμε ότι ορισμένα τέτοια ζευγάρια δεν αποφασίζουν να εγκατασταθούν σε κάποια χώρα που θα τους άρεσε γιατί δεν υπάρχει νομική ε, ασφάλεια, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες ε, προβλέψεις, δεν είναι εύκολο να υιοθετήσουν παιδιά, δεν αναγνωρίζεται η σχέση συμβίωσής τους σε ορισμένες ε, χώρες μέλη. Έχουμε λοιπόν δύο κανονισμούς και τονίζω ότι η άποψη των ειδικών ήταν ότι θα αρκούσε ένας κανονισμός, κανονισμός. Και εγώ συμφωνώ. Μόνο για πολιτικούς λόγους έχουμε τώρα δύο κανονισμούς. Γιατί ο κανονισμός για τις καταχωρημένες ε, σχέσεις συμβίωσης δεν ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούσε να περάσει. Αλλά τώρα οι ε, προοπτικές ε, είναι καλές. Εγώ ως φιλελεύθερη θέλω να προβλέπετε η δυνατότητα επιλογής δικαίου για αυτές τις καταχωρημένες ε, σχέσεις συμβίωσης. Περιλαμβάνεται τώρα στο κείμενο και ελπίζω κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να υπάρξει πλειοψηφία για το θέμα αυτό. Καλές είναι τώρα οι προοπτικές. Αυτό όμως σημαίνει ότι χρειάζονται πολλές διευκρινήσεις ε, και ε, ειδικέ ρήτρε για κάποια κράτη-μέλη ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαστήριά τους σε περιπτώσεις περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να αποφασίσουν. Δηλαδή, αν έχουμε δύο Γερμανούς με μια τέτοια σχέση που ζουν στην Πολωνία, τότε εάν χωρίσουν θα πρέπει για τα περιουσιακά στοιχεία να μπορέσουν να απευθυνθούν σε γερμανικές αρχές και εκεί να γίνει η διαδικασία. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά δυστυχώς ορισμένα πράγματα είναι πολιτικά ανέφικτα σε αυτή τη συγκυρία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τα κράτη-μέλη τα οποία είναι πρωτοπόρα, χώρες όπως η Σουηδία, γενικά οι σκανδιναβικές χώρες, για τα κράτη-μέλη αυτά. Δεν πάει αρκετά μακριά αυτή η πρόταση, ενώ χώρες όπως η Πολωνία, η Ιταλία θεωρούν ότι οι προτάσεις αυτές το παρακάνουν. Για να επιτευχθεί λοιπόν συμφωνία, επειδή υπάρχει η αρχή της ομοφωνίας, θα δούμε τι θα κάνουμε. Η Κυπριακή Προεδρία διοργάνωσε μια μεγάλη συνδιάσκεψη στην Κύπρο. Τώρα η Ιρλανδική Προεδρία δεν το θεωρεί βέβαια ως ε, πρωταρχική προτεραιότητα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό το θέμα. Θα κάνω μερικές συμβαστικές προτάσεις, ούτως ώστε οι χριστιανοδημοκράτες ε, στο Ευρωκοινοβούλιο και ορισμένοι που είναι ακόμη συντηρητικότεροι να μπορέσουν να βρουν κάποια σημεία συμφωνίας για να υπάρξει ευρεία ε, συνένεση για, τις δύο, ε, για τους δύο κανονισμούς ε, για τα περιουσιακά στοιχεία. Είμαστε στη φάση ακρόασης. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι για το θέμα της κληρονομίας Θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό έχουν προχωρήσει και τα κράτη-μέλη πριν πάρουμε θέση ως Κοινοβούλιο. Θα περιοριστώ σε αυτά και βεβαίως ε, αν θέλετε να μου θέσετε ερωτήσεις αλλά ήδη εξ ε, να με συγχωρήσετε αν δεν μπορέσω να παρευρεθώ μέχρι το τέλο τη συζήτηση. Ευχαριστώ τον ε, δόκτωρα Ντίρινγκ από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον οποίο θα ακούσουμε, ο οποίο θα μα εξηγήσει γιατί ε, αυτή η δυνατότητα επιλογής δικαίου είναι η μόνη συνταγματικά κατοχυρωμένη λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Θα ακούσουμε τώρα τις ε, αναλύσεις από δύο εμπειρογνώμονες. Πρώτα από τον κύριο καθηγητή Χες, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck του Λουξεμβούργου. Και θα δώσω αμέσως το λόγο. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα είναι ο κανονισμός για την κληρονομική διαδοχή. Δεν θα τα αναφέρω όλα τα βασικά, τα βασικά στοιχεία. Θα θέλω απλώς να αναφερθώ στις κατευθυντήρες γραμμές του κανονισμού και να επιχειρήσω να απαντήσω στο ερώτημα με, αυτές τις, ε, αυτόν τον κανονισμό λύνονται τα βασικά προβλήματα των πολιτών και να τονίσω μετά ποια είναι τα σημεία που δημιουργούν προβλήματα. Ο κανονισμός αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αποδοχή για εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής, καθώς και την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου. Διαβάζοντας τον τίτλο, καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια ευρεία προσπάθεια από πλευράς του Ευρωπαίου νομοθέτη για να λυθούν τα θέματα, τα κληρονομικά, τα διαμεθοριακά ως να τον ευρύτερα. Μέχρι τώρα δεν είχε ποτέ επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Είναι πραγματική πρωτοπόρα εργασία. Ένας ολόκληρος τομέας δικαίου για το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση, μέχρι ακόμη και τα πιστοποιητικά. Όλα αυτά τα θέματα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν. Οπότε δεν έχουμε κάποιο πρότυπο η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως κάνει πρωτοπόρα εργασία στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Χρειάζεται αυτή η προσπάθεια. Να επενθυμίσω μία υπόθεση. Είχα καλέσει, είχα τηλεφωνήσει σε ένα δικηγόρο. Έχω μία πελάτησα, της είπα, ε, του είπα, έχει πάρει μια μικρή δικηγορο εχω μια πελατησα ειπα του περίπου 200.000 ευρώ. Υπάρχει ένα μικρό σπίτι μεταξύ των περιοχικών στοιχείων, υπάρχει ένα μικρό σπίτι στη Γαλλία, στο Massif Central, στο κεντρικό οροπέδιο, 60.000 ευρώ κοστίζει περίπου. Μπορείτε να μου κάνετε μια γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Κληρονομικό Δίκαιο για να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Βεβαίω, είπε, αλλά το πρόβλημα του πενέφερε κ. Λέχνερ ήταν ότι η κληρονόμος ήταν ε, η Γερμανίδα για τα γαλλικά ακίνητα έπρεπε να εφαρμοστεί το γαλλικό δίκαιο. Έπρεπε λοιπόν, μια μικρή κληρονομιά να εκτελεστεί με βάση δύο διαφορετικά δίκαια. Και το ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς είναι τα πράγματα από πλευρά γερμανικού δικαίου. Δεύτερον, πώς θα κληρονομηθεί αυτό το ε, μικρό σπιτάκι και πώς θα μπορέσει να απολαύσει των δικαιωμάτων της ως κληρονόμος στη Γαλλία για αυτό το σπίτι, να πάρει λέει, τα κλειδιά και να το γράψει στο εκτιματολόγιο. Και σας είπα, το κόστος για την εμπειρογνωμοσύνη και για το δικηγόρο ήταν περίπου 10 με 15.000 ευρώ. Δεν ζητήσαμε τόσο πολλά, αλλά παρόλα αυτά. Ήδη ένα μεγάλο τμήμα της κληρονομιά έχει χαθεί. Πέρα από το χρόνο και τα άλλα προβλήματα. Ήταν πολύ περίπλοκη η ε, εκπόνηση αυτής της ε, γνωμοδότησης. Χρειάστηκαν εβδομάδε για να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται. Τι λέει τώρα αυτό ο νέο κανονισμό για την κληρονομιά. Φασίζεται σε τρει αρχέ. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είχαν βοηθήσει πολύ την κληρονόμο αυτή. Πρώτη αρχή. Να είναι το, η ίδια η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο. Δηλαδή, ήταν ε, γερμανικό δικαστήριο για την κληρονόμο. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί συνολικά να ε, εκτελεστεί αυτή η κληρονομιά με βάση το γερμανικό δίκαιο. Δεν θα εφαρμόζεται καθόλου το γαλλικό δίκαιο για τα γαλλικά ακίνητα. Αυτή είναι η δεύτερη αρχή. Δεύτερη αρχή. Ενότητα για την αντιμετώπιση της κληρονομία. Αυτό προτείνει και εγγυάται ο κανονισμός. Και η τρίτη πρόοδος ε, που απλώς επιφέρει ο κανονισμός να υπάρχει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο και η Γερμανίδα κληρονόμος μπορεί με αυτό το κληρονομητήριο να πάει στη Γαλλία για να μπορέσει να μπει στο σπίτι αυτό. Δηλαδή μείον 10-15 ευρώ έξοδα. Δεν είναι και λίγο. Παρ' όλα αυτά, κάθε κανονισμός, κάθε νέο μέσο, ιδίω άμα είναι εντελώ νέο και προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν έχουν επιληθεί μέχρι τώρα, υπάρχουν σημεία που μπορούμε να συζητήσουμε. Σημεία που όταν θα κάνουμε αποτίμηση του νομοθετήματος μπορούμε ενδεχομένως να τα ξαναδούμε. Να αναφέρω ορισμένα. Πρώτον, Ο κανονισμός μιλάει για ε, ίδια δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο. Οπότε αρμόδιο το δικαστήριο στην τελευταία συνήθη κατοικία, στην τελευταία συνήθη διανομή του κληρονομούντος. Και πού είναι αυτό. Είναι πολύ περίπλοκο να καθοριστεί. Μπορεί για κάποια άτομα που ε, ταξιδεύουν σε πολλές χώρες να είναι δυσχερές. Για παράδειγμα, εγώ ως διευθυντής του Max Planck ε, ε, Μένω στη Χαδελβέργη και δουλεύω πολύ συχνά στο Λουξεμβούργο. Αυτό δημιουργεί δυσχέρειε. Υπάρχει όμως άλλη λύση. Καλύτερη λύση. Ειλικρινά δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, με ανησυχεί, εάν και κατά πόσο η έννοια της συνήθους διανομής δεν θα προκαλέσει πολλές αντιδικίες. Ιδιαίτερα για θέματα αρμοδιότητας, δικαιοδοσίας. Σε περιπτώσεις που οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν για το ποιο δικαστήριο, και αυτό συμβαίνει συχνά, θα πρέπει να είναι αρμόδιο, για ποια δικαιοδοσία. Αλλά προβλέπει ο κανονισμός ότι τα μέρη θα πρέπει να κανονίσουν ποια θα είναι η δικαιοδοσία και παράλληλα ότι ο κληρονόμος μπορεί να πει, να έχει το δικαίωμα, θέλω να εφαρμοστεί το δίκαιο της χώρας προέλευσής μου. Και θα μπορούσαν λοιπόν όλοι οι ε, κληρονόμοι, αν συμφωνήσουν, εάν ε, αποβιώσει ε, ο διαθέτης στην Ισπανία, εάν συμφωνούν όλοι του οι κληρονόμοι, η κληρονομιά να γίνει αποδεκτή στη Φιλανδία. Αυτό βεβαίως, εάν δεν το πει ο ίδιος ο διαθέτης, ότι θα ήθελα να γίνει αυτό στη Φιλανδία. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Θα ήταν μια καλή λύση και αυτή. Αντίστροφα λοιπόν, εάν δεν έχει επιλέξει ο διαθέτης την ε, Φιλανδία, μπορούν οι κληρονόμοι όλοι μαζί να πούνε θέλουμε στην ε, Φιλανδία να γίνει η εκτέλεση. Η εκτέλεση. Αλλά μπορεί να αποφασίσουν και όχι στη Φιλανδία. Ορισμένοι μπορούν να πούνε είναι κάτι, καινούρια, κάτι καινούριο, δεν είναι όμως και απόλυτα καινούρια. Όμως στο σημείο αυτό θα ήθελα κάτι συγκεκριμένο που αρχικά το προέβλεπε η Κομισιόν, δηλαδή ότι τα δικαστήρια να μπορούν να βρουν όλα τα δικαστήρια που θα μπορούσαν να εμπλακούν τρόπο για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ε, ήδη υπάρχει αυτό για ορισμένες σχέσεις μεταξύ δικαστηρίων, αλλά για σχέσεις μεταξύ δικαστηρίων άλλων χωρών δεν ισχύει. Και αν δούμε τη λέει Κομισιόν, πιστεύω ότι θα καταλάβουμε ότι η απευθείας επαφή μεταξύ δικαστηρίων είναι βασικό θέμα της συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας στην Ευρώπη και αυτό λοιπόν ελπίζω στο μέλλον να γίνει όλο και περισσότερο να μπορεί να γίνεται αυτός ο διάλογος μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου. Ένα άλλο θέμα, για το οποίο δεν είμαι απόλυτα πεισμένος, ένα θέμα που ε, σχετίζεται και με αυτά που ακούσαμε σήμερα το πρωί, είναι η διατάξη του κανονισμού για, για θέματα αποδοχής ε, αποφάσεων. Εδώ ε, η πρόταση κανονισμού βασίζεται στην πρόταση Βρυξέλλες 1. Ναι, αυτές είναι οι διατάξεις, οι οποίες βεβαίως έχουν αποδείξει ότι είναι καλές και έχουν κάπως εκλεπτυνθεί. Αλλά είναι οι σωστές αυτές οι διατάξεις. Είναι σωστές σε αυτές τις περιπτώσεις αυτές οι διατάξεις. Διότι σε περιπτώσεις κληρονομιάς έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχει μια αντιδικία μεταξύ ε, δύο ατόμων αλλά δηλαδή στην, ε, στον κανονισμό Βρυξέλλες 1 υπάρχει πολλές φορές σαφή αντιδικία. Αλλά στι περιπτώσει ε, κληρονομιά υπάρχουν διαφορετικέ καταστάσει όπου μπλέκονται πολλοί κληρονόμοι και δεν είναι σαφέ ποιο είναι ενάγων, ποιο ενάγεται κτλ. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτέ οι καλύτερε διατάξει σε αυτόν τον τομέα. Θα είχα προτιμήσει, για παράδειγμα, ο κανονισμό για την αναγνώριση ο απλοποιημένος κανονισμός αναγνώρισης για τις περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας να έχει χρησιμοποιηθεί. Διότι η αφαιρεγγιότητα επίσης είναι περίπτωση όπου υπάρχουν ε, διαφορετικοί εμπλεκόμενοι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο κανονισμός είναι πολύ ε, κοντύτερα στις περιπτώσεις κληρονομίας από ότι είναι ο κανονισμός Βεξέλλας 1. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολη είναι η κωδικοποίηση των ε, θεμάτων αστικής δικαιοσύνης. Είναι πολύ διαφορετικές καταστάσεις και είναι δύσκολα να υπάρχει μια γενική αντιμετώπιση. Δύο περαιτέρω σημεία. Ο κανονισμός έχει ένα άλλο τμήμα και θα περάσω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες την αποδοχή και ε, έγκριση των εθνικών πιστοποιητικών κληρονομίας. Των εθνικών κληρονομητηρίων λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Το τελικό κείμενο του κανονισμού μιλάει για αποδοχή. Η γερμανική μετάφραση μιλάει για χρήση για απόδειξη και παρόμοιες χρήσεις. Τι σημαίνει αυτή η διατύπωση. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμή το θέμα αυτό. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λιγάκι μέχρι, τους, μέχρι η, η νομολογία να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η αρχή της αναγνώρισης εγγράφων. Πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν για ε, απόδειξη. Αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Κάποιο, Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο, ωστόσο, είναι μια πολύ καλή επιλογή. Συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Λέχνερ. Πρέπει να είναι απλά διατυπωμένο για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς είναι μόνο προαιρετικό. Και επειδή είναι νέο και προαιρετικό, δεν ξέρω αν πραγματικά θα αξιοποιηθεί. Θα το αξιοποιήσουμε μόνο εάν τα επόμενα χρόνια, μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός, Έχουμε ακόμη δύο χρόνια και. Εάν εμπλέξουμε όλους τους διαφερόμενους φορείς, ούτως ώστε να δεχθούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έντυπα. Βεβαίως πρέπει να μας βοηθήσουν και οι συμβολιογράφοι. Ευτυχώς έχουν ε, συμμετάσχει από την αρχή. Βλέπετε λοιπόν, ανέφερα κάποια κενά που υπάρχουν ακόμη, αλλά η βασική μου ε, εκτίμηση Υπάρχουν πολλά άλλα προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι από το 2015 η κατάσταση των ε, πολιτών σε τέτοιες περιπτώσεις διαμεθοριακών κληρονομιών θα βελτιωθεί αισθητά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τα, τις συνέπειες που έχουν οι καταχωρημένες ε, συμφωνίες συμβίωσης στις περιουσιακές σχέσεις των συντρόφων θα είναι το επόμενο θέμα, ε, το αντικείμενο της επόμενης ομιλίας. Θα μας μιλήσει αυτό ο Δ. Άλμπιν Daring από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερω για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για αυτά τα δύο θέματα. Και θα ήθελα να πω αυτής εξ αρχής ότι δεν θα καλύψω όλα τα ενδιαφέροντα θέματα και όλες τις πτυχές αυτών των δύο θεμάτων, αλλά θα επικεντρωθώ ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της δικής μου παρέμβασης. Ε, πέρυσι, τον Απρίλιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μία γνωμοδότηση σε σχέση με τον προτινόμενο κανονισμό που αφορά τις περιουσιακές συνέπειες των καταχωρημένων συμφωνιών συμβίωσης. Εξετάσαμε ιδιαίτερα τα σημεία που ε, επισήμανε η κυρία Τέιν από την αμική Επιτροπή. Ε, και για, τις, ε, ε, για, τα, για, τα, για τους συζύγους υπάρχει το άρθρο για, τα, για το γαμικό καθεστώς και τις περιεχθέσεις για, για τα σύμφωνα συμβίωσης δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής δικαίου όπως υπάρχει για τους συζύγους. Αναφέρεται όμως το άρθρο 15 ο νόμος, το δίκαιο του, της χώρας στην οποία έχουν καταχωρηθεί συμβάσεις και είναι ο μόνος εφαρμοστέος νόμος, το μόνο εφαρμοστέο δίκαιο. Ο ΦΡΑ, ο οργανισμός μας, ε, εξέδωσε τη γνωμάτευσή του τον Μάιο του 2012 για τις περιουσιακές συνέπειες των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης που δεν προβλέπουν επιλογή δικαίου, ενώ στην περίπτωση των γάμων οι σύζυγοι έχουν δικαίωμα επιλογής δικαίου που να διέπει τις περιουσιακές του σχέσεις. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων κανονισμών υπό το φως ε, ε, της ισότητας και του άρθρου 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης του άρθρου 21. Η ανάλυση μας λέει ότι θα πρέπει να βρούμε τις διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων κανονισμών. Από αυτή την άποψη να σημειώσουμε ότι η πρόταση που αφορά τις περιουσιακές ε, σχέσεις ε, δίνει στη συζύγους την επιλογή των, του εφαρμοστέου δικαίου για τις περιουσιακές του σχέσεις. Ιδιαίτερα ε, μπορούν να επιλέξουν το νομικό θεστός ε, της συνήθως της διαμονής τους ε, για τις περιουσιακές τους σχέσεις. Ως εκ τούτου, εξυπηρετείται και το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης τους, που είναι και το κυρίως θέμα της ε, με, της ε, μελέτης μας. Γιατί όμως το δικαίωμα αυτό επιλογής δικαίου που έχουν οι σύζυγοι να μην εξασφαλίζεται και για τους συντρόφους σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης υπάρχει διακριτική, διαφοροποιημένη μεταχείριση. Ε, οπότε φέρνει τα, τα ζευγάρια σε δυσμενή θέση σε σχέση με τα ζευγάρια διαφορετικού φύλου. Τα Ομοφυλόφιλα ζευγάρια που θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση του με ένα σύμφωνο συμβίωση δεν έχουν δυνατότητα επιλογή του δικαίου. Μόνο ένα εφαρμοστέο δίκαιο προβλέπεται για αυτού. Η προτινόμενη διαφοροποιημένη μεταχείριση, μάλιστα, είναι σημαντική και μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική διάκριση ορισμένων ομάδων. Οπότε το ερώτημα είναι, η διαφοροποιημένη αυτή μεταχείριση δικαιολογείται. Έχουμε τρία επιχειρήματα που προσφέρει η πρόταση. Αυτό που τονίζεται είναι η διαφορά μεταξύ των, των κανόνων των κρατών μελών που προβλέπουν ε, τις, τα, τις, σύμφωνα συμβίωσης. Παρόλο που σε κάποιο βαθμό υπάρχει μια κοινή έννοια του γάμου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό προς αρχές που τις διέπουν. Αυτό φαίνεται να ευνοεί την αντιμετώπιση των σχέσεων συμβίωση, υπό το πρίσμα του δικαίου που τις δημιούργησε, επιτρέποντα ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερε μεταβολέ σε σχέση με του γάμου. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα σχέδια κανονισμών δεν αφορούν τι νομοθετικέ διατάξει σχετικά με το γάμο και τι καταχωρημένε σχέσει συμβίωση, αλλά μόνο τα περιουσιακά δικαιώματα που συνδέονται με του θεσμού αυτού. Τώρα, όταν πρόκειται για καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, οι εθνικέ νομοθεσίε των κρατών μελών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Πολλά δικαιικά συστήματα στηρίζονται στην αρχή τη κοινή περιουσία των συζύγων, αλλά υπάρχουν επίση δίκαια που διέπονται από την αντίθετη αρχή, δηλαδή την αρχή τη περιουσιακή αυτοτέλεια. Δικαιολογημένα λοιπόν η πρόταση επισημαίνει τι δυσκολίε που προκύπτουν από τι σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των εφαρμοστέων κανόνων ουσιαστικού δικαίου προκειμένου να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα θέσπιση κοινού νομικού πλαισίου για τα περιουσιακά δικαιώματα των συζύγων. Ωστόσο, βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ίδιο ισχύει και υπέρ των καταχωρημένων συντρόφων. Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι ακριβώ οι διαφορέ μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών εκείνων των κρατών μελών που προβλέπουν τι καταχωρημένε σχέσει συμβίωση που δημιουργούν την ανάγκη θέσπιση συντονιστικού νομοθετικού μέσου και δίνουν ακόμη μεγαλύτερο βάρο στο ζήτημα τη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου. Δεύτερον, υποστηρίζεται ότι η απέτηση, οι περιουσιακές συνέπειε των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης να διέπονται πάντα από το δίκαιο του κράτους καταχώρησης βρίσκεται σε συμφωνία με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών που ρυθμίζουν τις καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης. Το δεύτερο επιχείρημα επισημαίνει το γεγονό ότι οι νομοθεσίε των κρατών μελών σχετικά με τι καταχωρημένε σχέσει συμβίωση δεν επιτρέπουν στου συντρόφου να επιλέξουν άλλο δίκαιο διαφορετικό από αυτό του κράτου καταχώρηση πρέπει καταρχά να υπενθυμίσουμε ότι η θέση του νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική από αυτή των νομοθετών των κρατών μελών. Ενώ η εθνική νομοθεσία στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αποσκοπεί στην αποτροπή συγκρούσεων δικαίου, τοποθετώντα τα εθνικά δικαιϊκά συστήματα σε μια διεθνή ανομή ο ρόλο τη νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες αξιώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως είναι η προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή στοιχεία που αναιρούν την υπόθεση ότι τα κράτη-μέλη αποκλείουν οποιαδήποτε δυνατότητα των καταχωρημένων συντρόφων να επιλέξουν καθεστώ διαφορετικό από αυτό του δικαίου του κράτου καταχώρηση. Στην Αυστρία, την Ολλανδία και τη Σουηδία οι καταχωρημένοι σύντροφοι έχουν τέτοια επιλογή, γι' αυτό και η γενική παρατήρηση ότι τα κράτη-μέλη δεν παρέχουν στου καταχωρημένου συντρόφου το δικαίωμα επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου συζητήματα σχετικά με τα περιουσιακά του δικαιώματα, φαίνεται να είναι λιγότερο κατάλληλη για να αποτελέσει τη βάση ενό ευρύτερου επιχειρήματο. Τρίτον, υπογραμμίζεται ότι δεν αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη τι καταχωρημένε σχέσει συμβίωση και ότι συνεπώ η έκταση Τη επιλογή δικαίου θα μπορούσε να μην είναι ίδια για έγκαμα ζευγάρια και για καταχωρημένου συντρόφου. Το επιχείρημα αυτό βασίζεται στο γεγονό ότι ενώ, ενώ τα κράτη-μέλη ρυθμίζουν με νόμο το γάμο, δεν σημαίνει το ίδιο με τι καταχωρημένε σχέσει συμβίωση. Αυτό είναι αληθέ και σημαίνει ότι για του καταχωρημένου συντρόφου, η δυνατότητα επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου περιορίζεται σε εκείνα τα κράτη-μέλη που διαθέτουν τέτοιου θεσμού. Ωστόσο, το γεγονό αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να στερηθούν ακόμη και μια τέτοια περιορισμένη επιλογή. Ο αναγκαστικό περιορισμό σε καθεστώτα που προβλέπουν την αναγνώριση των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωση δεν προσφέρεται ω επιχείρημα υπέρ τη αποστέρηση των καταχωρημένων συντρόφων, ακόμη και από το δικαίωμα επιλογή μεταξύ των υπολείπων ενόμων τάξεων. Οπότε ο Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέληξε στο συμπέρασμα στη γραμματότησή του ότι η αποστέρηση των καταχωρημένων συντρόφων από τη δυνατότητα επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου θα πετούσε επιχειρήματα που δεν μπορούν να, αντληθούν αντιληθούν από του λόγου που περιέχονται στην πρόταση. Συνεπώ, ο αποκλεισμό οποιασδήποτε δυνατότητα επιλογή δικαίου δεν φαίνεται να είναι σύμφωνο με την αρχή τη ισότητα του άρθρου 20 του χάρτη. Δεύτερον, η απαγόρευση των διακρίσεων στο άρθρο 21 του χάρτη θα απέκλειε μεταχείριση η οποία θα ευνοούσε τα παντρεμένα ζευγάρια, αλλά θα έθετε σε μια ανεκτική θέση τα άτομα τα οποία λόγω πολιτικής ή άλλης άποψης θεωρούν σημαντικό το να διάγουν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή με ένα μέγιστο βαθμό αυτονομίας και χωρίς κρατική παρέμβαση. Επίσης, δεδομένου ότι σε πολλά κράτη-μέλη ο θεσμός τη καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή για ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Μια τέτοια διαφοροποιημένη μεταχείριση θα ισοδυναμούσε σε, με έμεση διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Τερίν. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Θα ακούσουμε παρεμβάσεις, ερωτήσεις απευθυνόμενες προς τους ε, ομιλητές ή προς τους βουλευτές εδώ στο βήμα. Παρακαλώ να αναφέρετε το όνομά σας και να κάνετε μια σύντομη παρέμβαση. Ανοίχτε την καλοσύνη. Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση στα όσα υποθήκαν. Ο κ. Λένερ. Ευχαριστώ καθηγητά Χες, ευχαριστώ για τη θετική αποτίμηση. Όντως και εγώ προσωπικά και όλοι που συμμετέχαν, συμμετείχαν όπου υπήρχαν δυσχέρειες προσπάθησαμε ό,τι καλύτερο. Προσπαθήσαμε να χωρίσουμε τα επίμαχα θέματα ε, από, τα πιο, ε, από τα μη επίμαχα και ήταν δύσκολο να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Από πλευρά μου, οι, κανονισμοί για την ε, δικαιοδοσία είναι αποκλειστικοί. Ο Φινλανδός που ε, κληρονομεί κάτι στην Ισπανία μπορεί να κληρονομήσει στην Φιλανδία μόνο εάν ε, ε, ε, επιλέξει το δίκαιο της, της Φιλανδίας. Πρέπει λοιπόν να πω ότι ένας Γερμανός συνταξιούχος αποθάνει στη Μαγιόρκα και δεν έχει επιλέξει ο διαθέτης τη Γερμανία, τότε οι Γερμανοί ε, κληρονόμοι του πρέπει να επιλέξουν το ε, ισπανικό δίκαιο. Έτσι δεν είναι. Το ερώτημα λοιπόν ποιο είναι. Α, συγγνώμη, κάντε και μια παρατήρηση για τα εθνικά κληρονομητήρια. Αποκλείεται κατά τη γνώμη μου ότι μέσω του άρθρου 59 για την αναγνώριση εγγράφων είναι δυνατόν να μεταφερθεί η ισχύ ενός εθνικού κληρονομητηρίου πέραν των εθνικών συνόρων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται. Ε, βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ε, τράπεζες, από κάποιες αρχές σε μια άλλη χώρα έτσι για λόγους χρήσης. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα θα το αναγνωρίσουν. Θεωρείται λοιπόν ότι ο κανονισμός για την ε, δικαιοδοσία, για το ποιος θα εκδώσει το κληρονομητήριο διαφορετικά από το ότι βλέπετε την ε, εθελούσια δυνατότητα επιλογής δικαιοδοσίας. Τι κίνδυνος υπάρχει να υπάρχουν διαφορετικά κληρονομητήρια, διαφορετικά έντυπα που να οδηγούν σε διαφορετικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Και η Αλεξάνδρα θα ήθελε να πει κάτι από αυτού και θα απαντήσετε μαζί. Με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι ακόμη. το κλινομητήριο δημιουργεί, το ευρωπαϊκό κλινομητήριο δημιουργεί πρόβλημα στο κοινοβούλιο γιατί δεν υπάρχει σε διάφορες ε, χώρες. Ήταν δύσκολο σε χώρες όπου δεν υπάρχει, στη Γερμανία το ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήταν δύσκολο να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό το κλινομητήριο. Δεν καταλάβαιναν περί τίνος πρόκειται. Δεν κατάλαβαν τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το κλινομητήριο. Και αυτό ε, αντανακλάται και στα κείμενα. Ξέρετε ότι μια διαθήκη μπορεί να ανακαλυφθεί και 20 χρόνια μετά το θάνατο, άρα θα πρέπει να διορθωθεί το κλινομητήριο. Θα πρέπει μετά 25 χρόνια τώρα όλα να ξαναγίνουν. Αυτά μας λένε. Είναι πολύ δύσκολο. Οι βουλευτές που δεν γνωρίζουν αυτό το θεσμό να καταλάβουν τι επιπτώσεις έχει. Είναι ακόμη ασαφές ε, στο μυαλό πολλών για την δικαιοδοσία των δικαστηρίων επίσης. Για θέματα κληρονομικού, περιουσιακού και οικογενειακού δικαίου που είναι πολύ δυσχερείς είναι πιο δύσκολα ω τομεί από ότι είναι το δίκαιο των πωλήσεων από μια σύμβαση πωλήσεων είναι σκόπιμο τα δικαστήρια να εφαρμόζουν το δικό τους δίκαιο. Προσπαθήσαμε να το επιτύχουμε, διότι παρά όλη την δυνατότητα νομικής βοήθειας και όλα τα website είναι πολύ δύσκολο. Ιδίω για τους δικαστές ε, σε μικρές χώρες στην ε, Γερμανία έχουμε ειδικά δικαστήρια που ασχολούνται αποκλειστικά με την ε, εφαρμογή ξένων δικαίων, αλλά σε μικρές χώρες είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρετε αν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο το πορτογαλικό, το ουγγρικό δίκαιο κτλ. Με το τηλέφωνο δεν μπορεί να πάρει κανεί πληροφόρηση. Στόχος μας λοιπόν πρέπει να είναι ένας δικαστής στο μέτρο του δυνατό να χρησιμοποιεί το δικό του δίκαιο που το γνωρίζει. Και για τον κανονισμό για τα περιουσιακά στοιχεία Για παράδειγμα, ξέρετε ότι ε, οι απαιτήσει ε, συντάξεων ε, και αυτές συμμετέχουν στα περισσοκά στοιχεία, είναι τμήμα των περισσοκά στοιχείων, προσπαθήσαμε αυτά να τα, όλα αυτά να τα εξαιρέσουμε γιατί είναι πολύ ε, περίπλοκοι οι θεσμοί. Ακόμη και οι Αυστριακοί μας είπαν, κυρία Τάιν, καταλαβαίνουμε γερμανικά, αλλά αυτά τα θέματα παρακαλώ δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτές είναι συγκεκριμένες δυσχέρειες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για μια αρκετά γρήγορη απάντηση θα δώσω το λόγο στην κυρία. Μετά. Πολύ σύντομα. Ξέρω πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση, πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση των εθνικών συστημάτων και για τα περιουσιακά και συγκεκριμένα για τα κληρονομικά. Αντίστροφα, το Ευρωπαϊκό Κρονομητήριο είναι υπόδειγμα για το πώς μέσω νομοθεσίας μπορεί η Ένωση να ε, προκαλέσει μεταρρυθμίσεις και στα εθνικά δίκαια μέσω αυτής της ε, προσπάθειας. Εγώ θα ήθελα για την ε, διαμεθοριακή εξέταση ε, κληρονομικών διαφορών να εξαιρέσουμε ίσως τα κληρονομητήρια γιατί είναι περίπλοκη η κατάστασή τους. Αλλά δεν έχω πολλούς φόβους ότι θα υπάρξουν τρομερές διαφορές για τα θέματα της δικαιοδοσίας. Μπορεί να προκύψει. Η βασική μας όμως ιδέα είναι κυρίως να ε, εκτελούνται οι κληρονομίες από ένα δικαστήριο. Αλλά με βάση την πείρα μου, έχοντας παρατηρήσει το ξένο δίκαιο, έχω διαπιστώσει και κάτι που δεν, ε, δεν αρέσει πολλούς συναδέλφους που το λέω, θεωρώ ότι ορισμένες πορεί περίπλοκες ερωτήσεις δεν τίθενται καν για να μπορέσουν οι δικαστές να εφαρμόσουν ε, το δίκαιο που γνωρίζουν και για να καταλήξουν σε αποφάσεις. Αλλά υπάρχουν ερωτήματα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο που είναι σκόπιμο να αποφασίζονται τα θέματα δικαιοδοσίας και τα θέματα εφαρμοστέου δικαίου αφού πρώτα εξετάσουμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Βεβαίω είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνεται. Στο δίκαιο των προνομιών πάντα προσπαθεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι δύσκολο. Στο περιουσιακό ίσω να είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν είμαι όμω εμπειρογνώμων γι' αυτό. Εσεί, κυρία μου, πώ θέλετε να αντιδράσετε, να πείτε κάτι σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι μέλο τη ε, νομική επιτροπή αλλά ο συμπρόεδρος της ε, ομάδας για τα άτομα ε, LGBTT θα με ενδιαφέρουν οι προτάσεις σας. Τα άτομα λοιπόν ε, ομοφιλόφιλους, λεσβίες, διασεξουαλικά και μεταβατικά άτομα. Θεωρώ λοιπόν ότι τους, δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν και αυτό είναι κατά του άρθρου 22 της Χάρτας των Δικαιωμάτων. Ερώτημα ερώτημα και προς όλους. Όλοι, ξέρετε, παίρνουμε πολλά email που λένε ότι μέσω της ε, ε, ελεύθερης διακίνησης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβάλλει τους γάμους ομοφύλων σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ βέβαια θα έλεγα ε, όσο περισσότερη αρτότητα έχουν τα ζεύγη γκέι και λεσβιών το καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η νομική ε, πρόθεση. Εμείς θέλουμε να υπάρχει σίγουρα ελεύθερη διακίνηση για όλους. Ερώτημα λοιπόν. Τι νομικά επιχειρήματα εκτός από αυτά που ήδη αναφέρατε έχετε ούτως ώστε να καταστεί ακόμη σαφέστερο ότι στόχος μας είναι αυτή η αρχή της ελεύθερης διακίνησης που όλοι την έχουν αναγνωρίσει να μπορεί να εφαρμοστεί, να ισχύει ισότιμα και για τα ζεύγη γκέι και λεσβίων, είτε είναι παντρεμένοι, είτε αν έχουν σχέση συμβίωσης, παξ, οποιαδήποτε σχέση. Παρακαλώ, ε, δώστε μου επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι σίγουρα η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου αναγκαστικά περιορίζεται στα υπάρχοντα δίκαια, δηλαδή στα δίκαια των χωρών μελών που έχουν ε, στην ομοθεσία τους ε, το θεσμό των καταχωρημένων συμβάσεων, συμφωνιών συμβίωση. Δεν θα πρέπει να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη, να τα ξαναγκάσουμε να εφαρμόσουν ένα δίκαιο ή μια νομοθεσία που δεν αναγνωρίζει αυτά τα, αυτές τα σύμφωνα συμβίωσης. Γιατί μιλάμε για επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, όχι για το, την εφαρμογή του ίδιου ουσιαστικού δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντική αυτή η διαφοροποίηση. Μιλούμε επιλογή δικαίου μεταξύ νομοθεσιών που προβλέπουν αυτές οι καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης. Ε, πρόκειται για νομοθεσίες που έχουν εγκριθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτή είναι η βάση για το δικαίωμα της επιλογής. Τώρα, αν κληθούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση. Αν ένα ζευγάρι που μένει σε ένα κράτο μέλο ε, έχει το δικαίωμα να επιλέξει, είναι υποχρεωμένο να επιλέξει το δίκαιο της ε, χώρας διαμονής ε, σε περίπτωση που προβλέπει αυτό το δίκαιο στις καταχωρημένες σχέσεις δεν μπορώ να δω πως μια τέτοια επιλογή μπορεί να επηρεάσει άλλες χώρες που δεν προβλέπουν τέτοια δυνατότητα συμφώνου συμβίωσης για, τους, ε, για τα ζευγάρια που διαμένουν στο έδαφος τους. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Παρακαλώ. Πείτε μας το όνομά σας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την δυνατότητα που έχω να παρακολουθήσω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη. Είμαι μηχανικός πληροφορικής και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που συζητάμε. Τι γίνεται με την αναγνώριση ενός παιδιού που είναι, έχει γερμανική υπηκότητα, ενώ ο, ο πατέρας διαμένει στο Βέλγιο, για παράδειγμα. Η απόφαση του γερμανικού δικαστηρίου λέει ότι ο πατέρας καλείται να πληρώσει διατροφή. Έχει σταλεί η απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου στο Βέλγιο. Μέχρι ότου όμως αναγνωριστεί η απόφαση αυτή από το Βέλγιο, από τις βελγικές αρχές, και μέχρι ε, ότου προσπαθήσει ε, το Βέλγιο να ε, εκτελέσει την απόφαση του Γερμανικού Δικαστηρίου, θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα. Μερικέ φορέ και δύο χρόνια χρειάζονται για να περάσει το ποσό τη διατροφή στο λογαριασμό. Αν λοιπόν υπάρχει τέτοια κολλησιεργία, δεν έχουμε πραγματικά δικαιώματα. Ίσως θα πρέπει να προβλέψουμε μια διαδικασία που θα ε, επιταχύνει την πληρωμή αυτή από τον πατέρα προς το παιδί. Να γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Ε, ναι, βεβαίως, γι' αυτό έχουμε τον κανονισμό για διατροφή. Όπου αναφέρεται ότι κάθε κράτος μέλος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει μια κεντρική υπηρεσία όπου η μητέρα του παιδιού που ε, δικαιούται διατροφή πρέπει να μπορεί να βρει βοήθεια. Στη Γερμανία έχουμε κάνει ένα τέτοιο οργανισμό εδώ και ένα χρόνο. Δεν έχω ακούσει ε, διαμαρτυρίες από τη Γερμανία, διότι γνωρίζαμε τα προβλήματα αυτά. Γνωρίζαμε, δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε στην τύχη του τον γονιό που είναι υπεύθυνο για την ε, ανατροφή του παιδιού. Πρέπει να υπάρξουν διασυνοριακές ρυθμίσεις, πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες και καθήκον τους λοιπόν είναι των ε, κρατών μελών να υπάρξει ε, γρήγορη λύση. Πρώτη φορά ακούω ότι υπήρξε περίπτωση όπου καθυστερεί δύο χρόνια η διατροφή έχει αποφασιστεί αυτός ο κανονισμός ήδη από την προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Αυτός ο κανονισμός, καθώς και ο κανονισμός για το χωρισμό και οι κανονισμοί για τα προσωπικά στοιχεία, όλοι αυτοί οι κανονισμοί θα μας βοηθήσουν καθώς και οι κανονισμοί για την εκτέλεση αποφάσεων ε, στο εξωτερικό θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε τις προσπάθειές μας στο οικογενειακό δίκαιο. Αλλά φυσικά δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Ο, ο κανονισμός αυτός βεβαίως είναι ιδιαίτερα καινούριο. Πρέπει να δούμε πότε άρχισε να ισχύει. Και βέβαια κάποια κράτη-μέλη, παρά το ότι είναι κανονισμοί, δεν τα ε, μεταφέρουν, μεταφέρουν στην εθνική νομοθεσία με την ταχύτητα με την οποία θα έπρεπε. Είναι λυπηρό, αλλά έτσι είναι. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, διευκρινήσεις. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Αφορά ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο που αφορά την παρένθετη μητρότητα. Δίνω το λόγο στην κυρία Λονάς Μπρινέ για μια συγκριτική μελέτη στο θέμα αυτό. Έχετε το λόγο κυρία μου πατήστε το κουμπί για το μικρόφωνο σας. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν αυτή την προσωρινή έκθεση, ενδιάμεση έκθεση όσον αφορά μια μελέτη έγινε κατόπιν ε, ανάθεσης του Κοινοβουλίου για συγκριτική μελέτη των νομοθεσιών όσον αφορά την παρένθετη μητρότητα να αναφερθώ σε κάποια μεθοδολογικά στοιχεία να ξέρετε τι ακριβώς κάνει. Έχουμε 18 μέλη, κοινωνιολόγους και νομικούς στην ομάδα μας που α, ουσιαστικά εργαζόμαστε υπό τη διαχείριση του London School of Economic Enterprise. Α, για την ώρα έχουμε ερευνήσει την ομοθεσία και την ομολογία όλων των ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούσαμε ότι πρέπει να εξεταστούν ε, ήταν οι πιο σχετικές. Λοιπόν, για να μπω στην ουσία του προβλήματος, ε, όλοι διαβάζουν τον τύπο, ξέρουν το πρόβλημα, όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο αντιμετωπίζουν το θέμα της παρένθετης μητρότητας από όταν πήρε διεθνή χαρακτήρα και τα στήρα ζευγάρια αποφασίζουν να περάσουν τα σύνορα αυτά και να ψάξουν αλλού και όχι μόνο στη χώρα τους που απαγορεύεται να γίνει κάτι τέτοιο, δεν είναι καλά οργανωμένη αυτή η μέθοδος, ε, να αποκτήσουν ε, ένα παιδί που δεν μπορεί να εγκυμονήσει η σύζυγος, δεν έχουμε στοιχεία. Ε, είμαστε στο πρώτο στάδιο των μελετών, είναι δύσκολο να έχουμε ποσοτικά στοιχεία. Αυτά που δημοσιεύονται στα διάφορα έντυπα λένε ότι περίπου 500 με 600 παιδιά γεννώνται με αυτόν τον τρόπο. Τα μισά γεννώνται στη ΣΥΠΑ και τα άλλα μισά ε, στην Ινδία με αύξηση στην Ουκρανία. Αλλά αυτά τα στοιχεία κατά την άποψή μου είναι ατελή και εν μέρει ανακριβή. Γιατί έχουμε τόσα προβλήματα το πρώτο εμπόδιο όσον αφορά την παρέθετη μητρότητα, διότι υπάρχει έλλειψη ακριβών στοιχείων, ε, διότι τα ζευγάρια, τα στήρα ζευγάρια, από τη στιγμή περνάνε, περνάνε τα σύνορα για δύο βασικούς λόγους. Ε, δεν ξέρουμε ακριβώς λοιπόν, δεν έχουμε ποσοτικά στοιχεία από πλευρά Υπουργείων Δικαιοσύνης κάθε χώρας, διότι είτε οι γονείς δεν ζητούν να εγγραφούν τα ελιξερικές πράξεις γέννησης ε, στο εθνικό μητρό όταν έχει γεννηθεί ζουν παράνομα σε ένα κενό νομικό και αρκούνται καθημερινά στις ε, πράξεις του αστικού δικαίου του εξωτερικού. Και δεν υπάρχουν ε, έγκυρες πράξεις γέννησης στις χώρες στις οποίες διαμένουμε το παιδί τους. Αυτή είναι η πρώτη, πρώτος λόγος. Δηλαδή μένει αόρατη αυτή η πρακτική και ο άλλος λόγος για τον οποίο παραμένει τόσο αόρατη η πρακτική ε, είναι και εξή. Πολλές, ε, ε, πολλές πρεσβείες και ληξιαρχικές υπηρεσίες ανέχονται αυτό καθεστώ, καταχωρούν τι εξαιρετικέ πράξει γέννηση που χορηγούνται στο εξωτερικό ενό παιδιού που βγαίνει από αυτή τη διαδικασία της παρέθεση μητρότητα, σαν να το παιδί αυτό το απέκτησε η κανονική μητέρα, να έχει γεννήσει η μητέρα χωρίς την παρένθετη μητρότητα. Αυτό έχει γίνει στην, το είδαμε ότι γίνεται στην Ισπανία. Οι εκπρόσωποι μας στην Ισπανία το διαπίστωσαν αυτό. Επί μακρόν, λοιπόν υπήρξε μεγάλη ανοχή από πλευράς των ε, υπηρεσιών της Ισπανίας που ε, κατέγραφαν στη, στο ληξιαρχείο τις γεννήσεις που έλαμβαναν χώρα στο εξωτερικό ε, όχι ως αποτελέσματα παρένθετης μητρότητας ε, διότι βλέπουμε από τα στατιστικά στοιχεία μια μεγάλη ε, αύξηση γεννήσεων στην Καλιφόρνια από πλευρά Ισπανών υπηκόων. Και στη Γαλλία έχουμε άμεσες εγγραφές και δεν ξέρουμε πώς γεννήθηκε το παιδί, αν γεννήθηκε από την στήρα μητέρα ή όχι από τη μητέρα που έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και η σχέση με το προηγούμενο θέμα Όλες αυτές οι πρακτικές επιταχύνθηκαν από όταν νομιμοποιήθηκαν σε κάποιες χώρες, νομιμοποιήθηκαν οι σχέσεις ομοφιλοφίλων, ατόμο του ίδιου φίλου, είτε μέσω γάμος, είτε μέσω νομίμου καταχωρημένης συμβίωσης και μέσω της νομικής αυτής προσέγγισης τα ζευγάρια μπορούν να έχουν παιδιά ε, καταφεύγοντας την παρένθετη μητρότητα και σε κάποιες χώρες ε, ε ασκείται αυτή η πρακτική. Στην Ισπανία, ομοφυλόφιλα ζευγάρια που χρησιμοποιούν την παρένθετη μητρότητα στην Καλιφόρνια και αλλού, δεν υπάρχει δυνατότητα να εξακριβώσει κανείς. Υπάρχει άγνοια ε, και ανοχή από πλευρά των αρμοδίων αρχών όσον αφορά την καταχώρηση των γεννήσεων. Λοιπόν, αυτή η χρήση από ζευγάρια ομοφυλοφίλων τη παρένθετη μητρότητα κάνουν να κινείται, να αλλάζει η κατάσταση στην ε, νομοθεσία. Θα είδατε και από τον τύπο της Γαλλίας. Στην Ινδία αποφασίστηκε για πρώτη φορά να εθετηθούν κανόνες. Δεν ξέρω, κανονισμός, νόμος, οδηγία που απαγορεύει την παρένθετη μητρότητα για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Για τα άτομα του ιδίου φίλου έχουμε μία αποκριστάλλωση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την αναγνώριση των σχέσεων ατόμων του ίδιου φύλου. Στην μελέτη μας έχουμε μια αποκρισταλωση των προβληματων που εξετάζει κοινωνιολογικά στοιχεία. Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία μέσω ε, ερευνών σε διάφορες κλινικές στην Ευρώπη που εφαρμόζουν την πανέθετη μητρότητα στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις κάτω χώρες και στην ε, πρώτη αυτή κοινωνιολογική μελέτη θα έχουμε και ποσοτικά στοιχεία και ένα άλλο τμήμα που θα ασχολείται περισσότερα με τα κοινωνικά διακυβεύματα της πανέθετης μητρότητας και βλέπουμε τα γνωστά διακυβεύματα όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ, αφορούν ουσιαστικά την ελευθερία και την προστασία της γυναίκας που φέρει το εμβρίο, η ιατρική φροντίδα που έχει παρέθετη μητέρα και το παιδί και τα οικονομικά θέματα που ρυθμίζονται. Από την πρώτη μελέτη βλέπουμε ότι οι τιμές ε, διαφέρουν, ναι, δεν αμελείται το κόστος. 1500 ευρώ στην Ολλανδία και 50.000 ευρώ σε κάποια ελληνική κλινική στην οποία, την οποία επισκεφθήκαμε. Κοινωνιολογικά αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Προσπαθούμε να έχουμε αξιόπιστα ακριβή στοιχεία. Από νομική πλευρά είναι πιο εύκολα τα πράγματα, διότι έχουμε ακριβέστερα στοιχεία. Επιλέξαμε να εξετάσουμε τις πιο, κάποιες χώρες συγκεκριμένες στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες. στην τελική έκθεση θα υπάρξει ένας πίνακας που θα παρουσιάζει ποια είναι η κατάσταση όλων των χωρών, σε όλες τις χώρες και μετά θα επικεντρωθούμε επί κάποιων χωρών πιο σημαντικών. Γιατί πιο σημαντικέ, Διότι υπάρχει περισσότερη νομολογία, υπάρχει ένα πλαίσιο νομοθετικό που έχει ψηφιστεί ή που εκολάπτεται, εγκυμονείται, ε, συγχωρήστε το λογοπαίγνιο. Ε, αποφασίσαμε λοιπόν να εξετάσουμε και άλλε χώρε, εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, διότι μπορούν να θεωρηθούν μοντέλα για να προτείνουμε κάποια μέρα ένα κοινό μοντέλο, πρότυπο για την παρέθετη μητρότητα, αλλά για να κατανοήσουμε επίση πώ εμπνέονται οι χώρε η μία από την άλλη και πώ η Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, κατάφερε να έχει συγκρίσιμο καθεστώ με αυτό τη Νοτιού ε, Αφρική νομικά συστήματα πολύ κοντά στον αφάτη παρένθετη α, μητρότητα με πληρέστατο νομικό πλαίσιο. Ήταν ενδιαφέρον λοιπόν να βλέπουμε τι γίνεται και εκτός Ευρώπης, να δούμε και άλλα πρότυπα νομοθετικά που μας βοηθούν να εξετάσουμε λεπτομέρειες των διαφόρων μοντέλων των ευρωπαϊκών. Θα εξετάσουμε τι γίνεται και στο ρωσικό δίκαιο, διότι και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Ίσως είναι στους αντίποδες του μοντέλου που θα διαλέξουμε για την Ευρώπη, επιτρέπει την παρένθετη ε, μητρότητα εμπορικής βάσεως και όχι απλή ε, παρένθετη μητρότητα άνευ οικονομικής αποζημιώσεως. Ε, άρα είναι πολύ φιλελεύθερη προσέγγιση στην παρένθετη μητρότητα και το ίδιο θα εξετάσουμε και διαφορετικά μοντέλα, πιο φιλελεύθερα, πιο ανοιχτά, όπως της Καλιφόρνιας ή στο Illinois, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, στον υπόλοιπο χρόνο να σας περιγράψω ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία χώρα πέρα από την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, που προέβλεψε μέχρι τώρα ένα πλήρες πλαίσιο για την παρέθετη μητρότητα. Πλήρες πλαίσιο τι εννοώ. Ένα πλαίσιο όπου ελέγχεται, ελέγχονται οι συνθήκες για την παρέθετη μητρότητα ε, από πριν. Εγκρίνει ένας δικαστής τη συμφωνία που γίνεται και υπάρχει και ιατρικό πλαίσιο για την παρέθετη μητρότητα και για την τεχνητή γονιμοποίηση και υπάρχει ε, νομοθεσία ε, για μεταφορά ε, της κυδαιμονίας. Γιατί εκεί είναι σοβαρά τα δικηδεύματα. Για το αστικό δίκαιο μας ενδιαφέρει πολύ. Είναι το πιο σημαντικό στοιχείο αυτό. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που προσπάθησαν να το διοργανώσουν μόνο την ιατρική υπερίθαλψη μέσω προσανατολισμών ή κώδικα καλής πρακτικής ή κώδικα προσπάθησαν να διοργανώσουν την ιατρική πτυχή της προστασίας της μέρημνα για την παρένθετη μητρότητα στην τελική έκθεση θα παρουσιάσουμε την όλη κατάσταση για την Ολλανδία και για το Βέλγιο. Εν πάση περιπτώσει, εκτός της Ελλάδος όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν ένα κενό ή εν πάση περιπτώσει ελλείψεις, κενά, νομικά κενά όσον αφορά το οικογενειακό καθεστώς για τα παιδιά ε, και όλα τα νομικά συστήματα αναγνωρίζουν στο δικαστή ένα σημαντικότατο ρόλο διότι ο δικαστής σήμερα είναι εκείνος που θα πρέπει να παρέμβει για να ρυθμίσει το θέμα ε, για το να συνδέσει το παιδί με το, ε, το ζευγάρι, με τους γονείς, εκείνους που θα το μεγαλώσουν. Και δεν αφήνεται το παιδί προσκολλημένο στη μητέρα που το γέννησε και στο σύζυγό της ή τον σύντροφό της. όσον αφορά λοιπόν την παρέθυνη μητρότητα, βλέπουμε ότι ε, δεν παίρνει τα σύνορα. Στη Γαλλία, στη Ρουμανία ε, και σε άλλες χώρες προσπαθούν ε, κάπως να κάνουν πιο τους κανόνες περιοθεσίας προς όφελος του παιδιού ούτε ώστε νομικά με αξιόπιστο τρόπο να αντιμετωπίσει το θέμα. Να υπάρχει μια σταθερότητα. Να υπάρχουν αδιάλεκτοι δεσμοί μεταξύ του παιδιού με τους γονείς σε διεθνέ επίπεδο, όσον αφορά τη μητρότητα, όταν υπάρχει διέλευση συνόρων όπου η παρένθετη μητέρα είναι αλλοδαπή, εκεί οι τάσει είναι πολύ διαφορετικέ. Από τη στιγμή που υπάρχουν δημόσια τάξει, κρατικά διακυβεύματα, υπάρχει μεγαλύτερη αυστηρότητα πλευρά δικαστού. Ε, αναφέρομαι στο ποινικό δίκαιο και στο διοικητικό δίκαιο από τη στιγμή που υπάρχει εμπόριο παιδιών, πώληση παιδιών, οι δικαστές είναι πραγματικά παρόντες και επιβάλλουν ε, ποινές, όχι ποινικέ κυρώσεις, όχι πολύ μεγάλα ποσά, αλλά όμως ε, επιβάλλεται ποινή σε εκείνους που συμμετείχαν σε αυτό το εμπόριο του παιδιού και που πούλησαν το παιδί του σε κάποιο στήρο ζευγάρι. Από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων επίσης υπάρχει κίνηση όταν χορηγείται ένα ταξιδιωτικό έγγραφο, μια θεώρηση ταξιδιωτική για να μπορέσει ένα παιδί να επιστρέψει στη χώρα των γονιών του, ε, υπάρχουν δισταγμοί, προβλήματα, εντάσεις. Η Γερμανία είναι πολύ διστακτική στο να εκδίδει ταξιδιωτικά έγγραφα για να επιτρέψει στο παιδί να, ξανα, να επιστρέψει και να ζήσει με, τα, με τους γονείς στη Γερμανία. Είναι αβέβαιη και η κατάσταση και στη Γαλλία. Σε άλλες χώρες είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσον αφορά το αστικό δίκαιο, Εκεί υπάρχει μεγάλη διάκριση ε, σε όλες τις χώρες, διάκριση μεταξύ πατέρα και μητέρα του στήρου ζευγαριού. Υπάρχει μία, λόγω κανόνος, λόγω νομοθεσίας επιτρέπεται το παιδί να προσκοληθεί πιο εύκολα στον πατέρα ε, και στον πατέρα το βιολογικό. Είναι αρκετά εύκολο αυτό λαμβάνεται η ξεχή πράξη του εξωτερικού αναγνωρίζεται ή παράγονται αμέσως οι ανάλογες συνέπειες στη χώρα, στη χώρα που διαμένουν οι γονείς. Σε 90% των υποθέσεων ο πατέρας του στήρου ζευγαριού μπορεί να αναγνωρίσει την πατρότητά του όσον αφορά το παιδί στην Ολλανδία, Γερμανία, στο Βέλγιο πάντα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αναγνωρίζετε. Όμως αντίθετα υπάρχει μεγάλη αντίσταση, σχεδόν κοινή θέση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες που μπλοκάρουν την αναγνώριση της μητρότητα. Δηλαδή όλες οι ευρωπαϊκές χώρες συμμερίζονται αυτή την παράδοση. Είναι... Η, μητέρα είναι πάντα βέβαιη, είναι αυτή που γέννησε λέγανε οι Ρωμαίοι. Εκεί υπάρχει το κόλλημα το μεγαλύτερο, διότι όλες οι χώρες θεωρούν ότι αν η πράξη γέννησης περιέχει το όνομα της θύρας μητέρας, αυτή η πράξη δεν μπορεί να αναγνωριστεί στη χώρα στην οποία τις οποίες υπήκοοι είναι ε, διότι παραβιάζεται η νομοθεσία του κράτους. Όλη η δυσκολία συγκεντρώνεται στο πώς συνδέεται το παιδί με την μητέρα της τύρα. Βλέπουμε όμως, τη μη παρένθετη μητέρα, ε, είναι δουλειά για το δικαστή αυτή, που καλύπτει το κενό είδαμε σημαντική αλλαγή όσον αφορά ε, το πώς συνδέεται με την μητέρα το παιδί. Η Αυστρία και η Ρουμανία είναι χώρες όπου λαμβάνονται αποφάσεις από το δικαστή του αστικού δικαστηρίου και αποφάσεις λαμβάνονται εκεί με καινοτόμο τρόπο. Θεώρησαν ότι οι ληξιαρχές πράξεις γέννησης του εξωτερικού θα πρέπει να αναγνωρίζονται στην Αυστρία ή στη Ρουμανία και αμέσως ε, καθιερώνεται η σχέση του παιδιού με το στήρο ζευγάρι πατέρα και μητέρα. Είναι μια εξέλιξη ε, που ε, προωθήθηκε από τους δικαστές αυτές τις χώρες και βλέπουμε μια αργή εξέλιξη προς το ελληνικό μοντέλο. Μπορούμε να, έχουμε, να καταλήξουμε σε κοινέ αξίες από αυτή την ενδιάμεση την πρωταρχική έκθεση. Ε, φαίνεται ότι αυτό που απορρέει από την πρώτη βολιδοσκόπηση είναι ότι οι δικαστές θέλουν να μην υπάρχει αμοιβή. Είναι πάρα πολύ αυστηρή. Από τη στιγμή που πωλείται ένα παιδί, θέλουν να επιτρέψουν να μπει το παιδί να, στην οικογένεια, ενταχθεί στην οικογένεια των γονέων που το θέλησαν, υπό τον όλο που το παιδί δεν θεωρείται αγαθό στη διάθεση κάποιου, σαν ένα καταναλωτικό αγαθό. Δεν προχωρήσαμε πάρα πολύ στον όλο προβληματισμό. Εξετάζουμε οι ευρωπαϊκοί κανόνες σε τι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ σε αυτή την ανάλυση. Θα είναι η τελική ανάλυση, ο τελικός προβληματισμός του θέματος, αλλά βλέπουμε τελικά ότι προφανώς οι ευρωπαϊκοί κανόνες που ευνοούν τη μετακίνηση ακόμα και για ιατρική περίθαλψη ευνοούν την ελευθερία να μπορεί να πάει κανείς για περίθαλψη σε μια περίθαλψη που δεν υπάρχει ή δεν είναι αρκετά προχωρημένη στη χώρα που ζει κανείς και να μπορεί να πηγαίνει σε άλλη χώρα αν θα μπορούσαν να καλύψουν και την παρένθετη μητρότητα και αυτή η ελευθερία εντό του ευρωπαϊκού χώρου να μετακινείται κανεί, να μετακινηθεί το στυρό ζευγάρι, να πάει στην Ελλάδα, Φερρυπίν. Είναι μια δυνατότητα η οποία θα πρέπει να συζητηθεί. Για την ώρα λοιπόν, αυτή η ελευθερία της μετακίνησης ε, εμποδίζεται από τι εθνικές νομοθεσίες, ε, μάλλον καλύπτεται από τις νομοθεσίες. Από την Ελλάδα καλύπτεται, ατελώς καλύπτεται από τη Βρετανία, κάθε χώρα προσπαθεί στην δική του ένωμη τάξη να βάλει κάποιες ρήτες διαμονής ή υπηκότητας ή θεαγένειας λέγοντας ότι μόνοι οι γονείς που διαμένουν στην Βρετανία ή στην Ελλάδα μπορούν να καταφύγουν στην παρέθετη μητρότητα που πραγματοποιείται στις εν λόγω χώρες. Γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς χωρών που είναι πιο φιλελεύθερες από άλλες σε αυτό το τομέα να περιορίσουν τον αντίκτυπο που έχει η νομοθεσία τους. Για την ώρα αληθεύει ότι δεν έχουμε ακόμα κάποιες προτάσεις να σας κάνουμε σε αυτή τη φάση του προβληματισμού. Ποιο είναι το καθεστώς το που διέπει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ε, μαγειρεύουν κάπως την κατάσταση, βρίσκουν λύσεις οι δίκαστες. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει αβεβαιότητα στον αυτό το καθεστώς των παιδιών, ακραία βεβαιότητα αδυναμία να προβλέψει κανεί από τον νόμο τι γίνεται. Τεράστια αβεβαιότηση υπάρχει σε αυτόν τον τομέα και σήμερα το πρωί ο Υπουργό Δικαιοσύνη της Ιρλανδίας εξέφρασε τον προβληματισμό του για αυτή την ανασφάλεια και επέμεινε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνε αξιόπιστοι να μπορούν το καλύπτουν αυτό. Και όσον αφορά την παρέθετη μητρότητα, ε, πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχόλια, απορίες για το θέμα της παρένθετης μητρότητα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Γιώνας Γκένεσον και είμαι μέλος της Σουηδικής Βουλής. Ήταν ε, καταπληκτική η παρουσίαση της κυρίας Μπρουνέτ και την ευχαριστώ θερμά γιατί πραγματικά ε, έθεσε το δάκτυλο επί των ήλων, γιατί αλλάζουν ε, οι κοινωνίες μας, αλλάζει η νοοτροπία, βελτιώνεται η στάση απέναντι στους ομοφιλόφιλους και δημιουργείται και η δυνατότητα να αποκτήσουν απογόνους μέσω της παρέθετης μητρότητας. Σημαντικές εξελίξεις λοιπόν και οι περισσότερες χώρες που επιτρέπουν τη διαθεσία από ζευγάρια ίδιου φύλου Ε, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Είναι πολύ θετική αυτή η νέα δυνατότητα που διαφαίνεται, γιατί δίνει την ευκαιρία και σε συντρόφους του ίδιου φίλου να γίνουν γονείς. Και ε, βέβαια, πολλές φορές, παρόλο που υπάρχει θεωρητική νομική δυνατότητα υιοθεσίας για τέτοια ζευγάρια, δεν την ασκούν και στην πράξη. Πάντως, για τις παρέθετες μητέρες, θα πρέπει να δούμε τι άλλοι δρόμοι υπάρχουν, τι άλλες λύσεις μπορούμε να αναζητήσουμε για να υπερκεράσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε πραγματικά την ευκαιρία ε, στους ε, ανθρώπους που το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους να γίνουν γονείς. Όπως ε, και με την υιοθεσία, να διευκολύνουμε την υιοθεσία σε περίπτωση που προσκρούει είτε σε νομικά προβλήματα είτε σε κοινωνικά. Υπάρχει και ένα άλλο αλληλένδετο θέμα. Δηλαδή ένα θέμα που συνδέεται με τη δυνατότητα των συντρόφων του ίδιου φίλου να αποκτήσουν οικογένεια. Είναι το θέμα της μητρότητας, ιδιαίτερα ε, σε ζευγάρια γυναικών γιατί υπάρχει δυνατότητα στις ε, λεσβείες μητέρες με τεχνική γονιμοποίηση να αποκτήσουν παιδί, αλλά τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται στη Σουηδία. Στη Δανία όμως είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Γιατί δεν χρειάζεται κανείς ε, να γεννήσει ένα παιδί για να το αισθανθεί δικό του παιδί. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν αυτή τη σχέση. Για να μην ε, αισθανθεί το παιδί απομονωμένο ή περιθωριπημένο από τον άλλο σύντροφο που δεν είναι η βιολογική του μητέρα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν πρώτα απ' όλα τα συμφέροντα του παιδιού και αυτό και στα πλαίσια τη παρέθετη μητρότητα. Σα ευχαριστώ. Θέλει άλλο κανεί το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ράσμασον από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ευχαριστώ την κυρία Λοράς Πρινέτ για την παρουσίασή της. Και θα ήθελα να ρωτήσω μήπως ε, οικειοθελώς ε, μας αποκρύψετε ένα θέμα βασικό, που είναι το θέμα του κατά πόσο είναι αποδεκτή αυτή η παρέθετη μητρότητα. Γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, ε, πολύ ευαίσθητα για τους πολίτες και τις κοινωνίες μας. Ή το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο στόχος της υποβοηθούμενης τεκνοποίησης. Ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να διορθωθούν κάποια ιατρικά προβλήματα ή μήπως ε, θέλουμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη που αισθάνονται μερικοί να αποκτήσουν παιδί, την επιθυμία. Γιατί μερικοί, για, όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά για άλλους λόγους, για παράδειγμα ομοφυλόφιλα ζευγάρια ή γυναίκες που, έχουν, ε, που βρίσκονται στην ημινόπαυση και παρόλα αυτά θέλουν να, να υποφεληθούν από την ενότητα υποβοηθούμενης ε, αναπαραγωγής ή από την παρέθετη μητρότητα. Μήπως λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμο ή βιώσιμο ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σχέδιο και κατά πόσο θα το ε, αγκαλιάσει η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρχει μια τέτοια κοινωνία των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω πάντως ότι ό,τι λύση και βρεθεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις εθνικές ευαισθησίες. Δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό ή δυνατό να καταλήξουμε από αυτήν την άποψη σε κοινού κανόνε πανευρωπαϊκούς δηλαδή, για τα ευαίσθητα αυτά θέματα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπρουνέτ, παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε. Μπορώ να απαντήσω ταυτόχρονα και στις δύο ερωτήσει γιατί επικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό. Τώρα, γιατί καταρχήν η παρένθετη μετρότητα είναι ένα μέτρο υποβοηθούμενης ιατρικά αναπαραγωγής. Δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το αντικείμενο της μελέτης της δικής μας, γιατί δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ούτε τον εθνικό ε, νομοθέτη, ούτε τον ευρωπαϊκό νομοθέτη. Είναι θέμα κοινωνιολογίας του δικαίου, δηλαδή οι πρακτικές αυτές υπάρχουν σε όλες τις χώρες σήμερα. Και το διαπιστώσαμε κάνοντας μια επισκόπηση και της νομολογίας. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα και το θέμα είναι να λύσουμε αυτά τα προβλήματα Ιδιαίτερα το θέμα του καθεστώτος που ισχύει για το παιδί. Και αυτό ήταν το αντικείμενο της μελέτης. Είδαμε ότι τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Μερικές φορές ε, αυτοσχεδιάζουν οι δικαστές και ε, καταφεύγουν σε διάφορα ευρήματα για να συνδέσουν το παιδί με τους γονείς. Ενώ ο εθνικός ή ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, μπορούν να καταλήξουν σε εθνικούς ή σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε τη συζήτηση επεκτείνοντάς την και στην κοινωνία των πολιτών. Μάλιστα στη Γαλλία επιβάλλει στην περίπτωση αυτή η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και αυτό ισχύει από το 2011. Τώρα για να αναφερθώ σε ένα πιο κοινικό ερώτημα που θέσατε. Το κατά πόσο δηλαδή θα μπορούσαμε να προτείνουμε, γιατί τονίσατε το ότι η παρέθετη μητρότητα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις από τότε που επιτρέπεται στα ζευγάρια του ίδιου φύλου να χρησιμοποιήσουν τέτοια πρακτική για να γίνουν γονεί. Ή αν θα μπορούσαμε να προσανατολιστούμε προ την ε, υιοθεσία. Να αφήσουμε κατά μέρο την παρέτητη μητρότητα και να επικεντρωθούμε μόνο στην υιοθεσία. Ε, διευκολύνοντας Διευκολύνοντα την υιοθεσία από τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Αλλά για την υιοθεσία υπάρχουν, ε, υπάρχει πληθώρα κειμένων και διατάξεων. Αλλά δεν υπάρχουν αρκετά παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Γνωρίζω ότι στη Γαλλία 30.000 ζευγάρια περιμένουν σε λίστα αναμονή για να υιοθετήσουν παιδί. Πέρυσι μόνο είχαμε 1.500 ζευγάρια. Ναι, μπορούμε να διευκολύνουμε ή να ε, ευνοήσουμε την ε, υιοθεσία το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει, αρκετά προσφορά, δεν υπάρχει προσφορά, δεν υπάρχουν παιδιά προς υιοθεσία. Γιατί οι χώρες ε, που προηγουμένως ήταν προμήθευαν κατά κάποιο τρόπο, ήταν πηγή για παιδιά προς υιοθεσία, τώρα ε, ενισχύουν ε, τον άλλο δρόμο να παραμείνουν τα παιδιά με τις βιολογικές τους μητέρες. Δεν ευνοούν την υιοθεσία. Οπότε μας μένει η παρέθετη μητρότητα και σας παραπέμπω εδώ και στην ενδιαφέρουσα νομολογία του ΔΕΚ για το θέμα αυτό. Πάντως, ακόμη και αν σκεφτούμε το θέμα της υιοθεσία και αφήσουμε ανοιχτό το θέμα και της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της υιοθεσία. και το θέμα είναι ότι αν δεν μιλήσουμε για την παρέθτη μητρότητα θα, προβλέπ, θεσπίσουμε πολύ σημαντική διάκριση μεταξύ αδρών και γυναικών γιατί έχουμε κάποιες πολύ πιο φιλελεύθερες νομοθεσίες που αναγνωρίζουν τις ε, οικογένειες ε, ιδίου φύλου και έχουμε την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία που είναι πιο φιλελεύθερες που επιτρέπουν σε ζευγάρια γυναικών να χρησιμοποιήσουν την υποβοηθούμενη ε, ιατρικά αναπαραγωγή αλλά οι ίδιες αυτές τις χώρες δεν προτείνουν τίποτα για τους άντρες, για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια ανδρών. Οπότε ανοίγουμε πολύ περισσότερο τη διαδικασία της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και διευρύνουμε τους καρόνες πρόσβασης ώστε ε, να μπορούν τα ζευγάρια δύο φίλου εφόσον είναι γυναίκες να έχουν τέτοια πρόσβαση αλλά τι θα γίνει με τους άνδρες ε, που ε, είναι μαζί, είναι σε τέτοιες σχέσεις ομοφιλόφιλες. Για αυτούς υπάρχει μόνο η παρέθετη μητρότητα ως λύση. Και ε, υπάρχει η δυνατότητα από το 2005 ε, η Συμφωνία, Σύμβασης, ε, η Συμφωνία Συμβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατα προβλέπεται δυνατότητα και παρένθεση μητρότητας ε, για τα ζευγάρια ίδιου φύλου. Είναι μια εξέλιξη που είναι δύσκολο να την αναχαιτήσουμε, πιστεύω, δεδομένες στις ραγδαίες της ΠΕΛΕ τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Εδώ θα έχουμε την Σεσίλια Βίξτρομ, που είναι η μοναδική εκπρόσωπος εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Και μετά θα ακούσουμε τον ε, Εφέτη από τη Λισαβόνα, τον κύριο Κάρλος Τεμέλο Μαρίνιο. Merci. Merci. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχάς ζητώ συγγνώμη για την απουσία της Κέρ Παρβανόβα και του κυρίου Λόπες. Θα θέλανε πάρα πολύ να είναι εδώ, παρόντες. Έπρεπε να κυρώσουν όμως λόγω ασθενείας. πρόσφατα ασθένησαν. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ όμως και μπορώ να συζητήσω μαζί σας το το αυτό νομικό θέμα, το κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση, για τα μέτρα προστασίας αστικά ζητήματα, δεν είναι πολύ σεξι σαν θέμα, είναι όμως. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες η ε, θέσπιση ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τα δικαιώματα των θυμάτων θα εξακολουθεί να προσφέρει σε όλα τα θύματα εγκληματικών ενεργειών ανεξάρτητα από την υπηκότητά τους ή που διεπράχθη το έγκλημα την αναγνώριση και την ευρύτερη δυνατή προστασία σε όλη την επικράτεια της ε, Ένωσης. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η πρόταση προέρχεται από τις διατάξεις της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας ε, που εκάλυπτε αρχικά όλο το φάσμα των μέτρων προστασίας που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη ανεξάρτητα από την αρχή αν είναι ε, του ποινικού ε, τομέα ή του αστικού τομέα η αρχή που εξέδωσε αυτό το ένταλμα. Ε, είδαμε τα σχόλια των διαφόρων, κρατικό, διαφόρων ε, κρατών ε, πώς αντιμετωπιζόταν αυτά τα θέματα και γι' αυτό θέλαμε να έχουμε ξεχωριστό μηχανισμό αναγνώρισης για την αστική προστασία και τα εντάλματα για την αστική προστασία και ο συνδυασμένη, η συνδυασμένη εφαρμογή των δύο μέσων ποινικό μέσο και αστικό μέσο θα επιτρέπει στα άτομα τα οποία καλύπτονται το ένταλμα προστασίας να κινούνται ελεύθερα και ασφαλώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 των συνθήκων μας. Η συνεισφορά μας όσον αφορά το κύμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεπνέεται από το βασικό στόχο. Θέλαμε γρήγορη και απλή αναγνώριση και όπου ήταν δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας, να εκτελούνται. Για να πετύχουμε το στόχο μας, κάναμε βασικές προτάσεις ε, που συμπεριλήφθησαν στο κείμενο. Στι τροπολογίε τροποποίηση του αρχικού κειμένου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέψαμε στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν και αυτομάτω να εκτελούν, εφαρμόζουν το ένταλμα αυτό που εκδίδεται από άλλο κράτο μέλο κατόπιν παρουσίαση ενό πιστοποιητικού που προέρχεται από το αρχικό κράτο μέλο. Πιστεύουμε ότι αυτό θα παράσχει μεγαλύτερη προστασία για πιθανά θύματα. Η διοικητική διαδικασία θα γίνει απλούστερη και θα εξασφαλίζεται η προστασία αυτών των ανθρώπων οπουδήποτε, οποτεδήποτε ταξιδεύουν και μετακινούνται προς ένα άλλο κράτος μέλος. Στην πρότασή μας επίσης προτείναμε να υπάρχει μια βάση δεδομένων, να δημιουργηθεί βάση δεδομένων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μέτρα προστασίας και τα διάφορα πιστοποιητικά που εκδίδονται. Ε, πιστεύουμε ότι έτσι οι, ε, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να δράσουν γρήγορα θα έχουν πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες και το τρόπο εξασφαλίζουν αποτελεσματική ταχεία διασυνοριακή προστασία κατά τυχών απειλών. Και τα προστατευόμενα άτομα που δεν ομιλούν την γλώσσα ε, στα πλαίσια των διαδικασιών που αφορούν τα μέτρα προστασίας θα, σε δικαστικές διαδικασίες κλπ. θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διερμηνία και σε μετάφραση όλες οι πληροφορίες και όλη αυτή η νομική βοήθεια που παρέχεται στο προστατευόμενο άτομο θα πρέπει να προσαρμόζεται και στις ατομικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου και θα πρέπει η μορφή που του παρέχονται οι πληροφορίες να είναι εύληπτη. Για να μειώσουμε περαιτέρω τα διοικητικά βήματα που απαιτούνται, συμφωνούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει τυποποιημένος πίνακας, τυποποιημένη μορφή εντύπου, πολύγλωση, άρα να αποφεύγεται η ανάγκη μετάφρασης και να επιταχύνεται η αναγνώριση. Πιστεύω λοιπόν, αντικαθιστώντας τους δύο εμπειρογνώμονες συναδεφέρθους μου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, αυτά είχα να πω και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κάλλος Δεμέλο Μαρίνιο, τον εμπειρογνώμονα το λόγο, που είναι δικαστής στο εφετείο της Λισαβόνας, θα ήθελα να σε ενημερώσω περί των διαδικασιών για την έγκριση αυτού του μέσου του εργαλείου. Τώρα, σε αυτή τη φάση, ετοιμάζουμε το δεύτερο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με όλα τα θεσμικά όργανα και ελπίζουμε βεβαίως να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, κάτι που ταιριάζει και με τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Έτσι νομίζω ότι σκιαγράφησα τα βασικά χαρακτηριστικά της ε, πρότασης και βεβαίως με τα χαράς να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλια. Αμέσως θα δώσω το λόγο στον κύριο δικαστή Καλησπέρα σα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ και σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι σίγουρος ότι ο κανονισμό θα είναι πολύ θελκτικός, πολύ σεξι και θα είναι και πολύ χρήσιμο γιατί αγγίζουμε εδώ την καρδιά μιας πολύ σημαντική ανάγκης των Ευρωπαίων πολιτών. Εγώ παρακολουθώ αυτόν τον κανονισμό από τα σπαργανά του και θυμάμαι ότι το 2003, το Σεπτέμβριο, ήμουνα στην Ιταλία και εκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας και ο κύριος Βιτορίνο, επίτροπος ε, για θέματα δικαιοσύνης, ε, ήρθε για να παρουσιάσει μέσα σε ένα σεμινάριο τριήμερο τον κανονισμό. Είπε ο υπουργό ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και ότι ο κανονισμός θα έφερνε τέρμα ε, σε μια κατάσταση στην Ευρώπη. Βέβαια, οι ανακοινώσεις αυτές δεν επαληθεύθηκαν. Τελικά το πιο σημαντικό πράγμα του κανονισμού έμεινε πίσω. Ήταν ε, ο κανονισμός του 2011 ε, 0130 ε, και από ό,τι ξέρω η πρώτη φορά είναι που καταπεί σε πλήρως τη διαδικασία αναγνώρισης και τον εκτελεστήριο τίτλο, τον, το εξεκουάτορ, σε δύο σε δύο ε, περιπτώσεις. Οι χώρες δεν ε, ε, έκαναν αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Και ο κανονισμός αυτός ήταν η έμπνευση και για ε, την, ε, το ένταλμα εκτέλεσης ή την, την εντολή για την πληρωμή. Πολλοί κανονισμοί και πολλές οδηγίες μετά τον ε, κανονισμό αυτό για την αμοιβή αναγνώριση μέτρων προστασία εμπνεύστηκαν από αυτόν. Και αν είχαμε άμεση επικοινωνία μεταξύ των δικαστών, δημιουργούμε ουσιαστικά τα θεμέλια της, του κοινού συστήματος απονομής δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Και ο κανονισμός αυτός έκανε αυτό που ήταν προφανές αλλά που έλειπε μέχρι τώρα. Δηλαδή, ε, προσπάθησε να ε, καταργήσει, να, να υποκαταστήσει αυτό το κενό της κατάργησης της αμοιβές αναγνώρισης στο μέτρο προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Καλύτερη, λοιπόν αυτό το κενό της ε, αναγνώρισης αυτών των μέτρων σε αστικές υποθέσεις είναι σαφές ότι μόνο με ένα οριζόντιο πλέγμα κανόνων μπορούμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο μας στόχο, να επιτρέψουμε δηλαδή τους δικαιούχους αυτών των μέτρων προστασίας ε, ε, και το δικαίωμά τους να μετα... μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Αλλιώς θα τους καταδικάζαμε σε μια κινητοποίηση, αν δεν υπήρχε αυτή η αμοιβή αναγνώριση. Αυτό το σχέδιο κανονισμού λοιπόν έχει, ενέχει το δυναμικό να δώσει ε, δικαίωμα μετακίνησης ε, ανθρώπων που βρίσκονται υπό απειλή, που απειλούνται με τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος. Και επίσης η διασυνοριακή προστασία μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα και στις δίκες γιατί επιτρέπει ελεύθερη πραγματικά και σωστή άσκηση των δικονομικών δικαιωμάτων. Μπορεί ε, να έχει και αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τη διάπραξη εγκλήματος και ως ε, ε, παρενέργεια μπορεί να έχει θετική παρενέργεια την σωστή ε, συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Μπορεί να μην είναι σεξι λοιπόν ο κανονισμό, αλλά είναι πολύ σημαντικός. Και οι αστικές υποθέσεις ε, αποφελούνται ιδιαίτερα από τον κανονισμό γιατί γίνονται ελαφρύτερες, ταχύτερε και πιο αυτόνομες. Τα μέτρα αυτά, μάλιστα, εκδίδονται από πολιτικά δικαστήρια, αστικά δικαστήρια και ουσιαστικά περιορίζουν κάποιον ε, από συγκεκριμένη δραστηριότητα ή τη χρήση ενός χώρου. Και μάλιστα τέτοιε, τέτοιες απαγορεύσεις μπορούν να αφορούν συγκεκριμένη συμπεριφορά ή την ε, χρήση ενός κοινού χώρου, ενός σπιτιού για παράδειγμα, μιας οικίας. Σε μία μελέτη που έγινε πριν την εκπόνηση αυτού του εγγράφου αναφέρεται ότι πολλά κρατημέλη ήδη έχουν κάποια εσωτερικά μέτρα προστασίας για αστικές υποθέσεις. Κάτι που καθιστά ακόμη μεγαλύτερη την ανάγκη να θεσπιστούν μέτρα για την διασυνοριακή αναγνώριση και εκτέλεση των τέτοιων αποφάσεων μέτρων προστασίας. Ο προτινόμενος κανονισμός εντάσσεται σε ένα πακέτο εγγράφων που δημοσιεύθηκε το 2011, περιλάβανε και την ανακοίνωση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων, μια πρόταση οδηγίας για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα των θυμάτων, ένα ψήφισμα του Συμβουλίου για ένα οδικό χάρτη προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων, ιδιαίτερα σε ποινικέ δίκες. Και έχουμε και αυτή την πρόταση που ουσιαστικά συμπληρώνει τα προηγούμενα νομοθετικά κείμενα και θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση στο υπόλοιπο πρόβλημα, δηλαδή την παρέμβαση των δικαστηρίων σε αστικές υποθέσεις και την έκδοση απόφασης τους ε, για μέτρα προστασίας και την αναγνώριση αυτών των μέτρων προστασίας σε άλλες χώρες προκειμένου να μπορούν οι πολίτες που είναι δικαιούχοι αυτό το μέτρο να μετακινούνται ελεύθερα. Ποιοι είναι οι στόχοι. Ο βασικός στόχος ε, της ε, θέσπισης ενός τέτοιου κανονισμού είναι να γλιτώσει τον κόσμο από δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες. Γιατί εδώ το, ο χρόνος είναι χρήμα και πολύ σημαντικός. Μιλούμε για την προστασία θυμάτων που ανα πάσα στιγμή μπορούν να αποτελέσουν ε, στόχο μια εγκληματική ενέργεια. Οπότε είναι θεμελιώδη σημασία να κερδίσουμε χρόνο εδώ. Τώρα, πώ η πρόταση αυτή κερδίζει χρόνο, πώς επισπεύδει τις διαδικασίες. Μα δημιουργεί ένα πιστοποιητικό, ένα δημόσιο έγγραφο που είναι κοινό και που εκπληρώνει την ανάγκη της ελεύθερης κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων. Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που μπορεί να εφαρμοστεί, να εκτελεστεί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπορεί να εξασφαλίσει την άμεση προστασία του θύματος οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν, αποτελεί την καρδιά της πρότασης αυτό το πιστοποιητικό. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο του κανονισμού αυτού είναι η δυνατότητα επέκταση των μέτρων σε χώρες που δεν εφαρμόζουν τέτοια μέτρα, που δεν διαθέτουν τέτοια μέτρα. Για παράδειγμα, στη δική μου την πατρίδα, την Πορτογαλία, υπάρχει ένα καλό σύστημα, τουλάχιστον θεωρητικά, για ηλεκτρονικά βραχιόλια που ε, εξασφαλίζουν, την παρακολούθηση των υπόπτων για παρενόχληση ή των υπόπτων διάπραξη εγκληματικής ε, ε ενέργειας. Αν δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα στο Βέλιο, για παράδειγμα, με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το ε, δυνητικό θύμα μπορεί να ζητήσει από το Βέλγιο να εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα, προκειμένου να εκτελεστεί η απόφαση του Πορτογαλικού Δικαστηρίου, που περιλαμβάνει τέτοια μέτρα, του ηλεκτρονικού βραχιολίου για παράδειγμα. Βέβαια δεν έχουμε μια συμμετρική πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε ομοιομορφία. Μερικές χώρες δεν έχουν απαντήσεις ε, ε, στις ανάγκες των θυμάτων για προστασία. Οπότε αυτή η πρόταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η τελική λύση, η οριστική λύση. Ούτε θα είναι η κατάληξη της διαδικασίας, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παρόμοιες δομές και μέτρα για την προστασία των θυμάτων σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κοινέ δράσεις ώστε να απολαμβάνουν ίδιας προστασίας οι πολίτες παντού. Πάντως η πρόταση αυτή δίνει μία απάντηση σε ένα θεμελιώδες ζήτημα στην ανάγκη ε, ε, εκτέλεσης, ε, διασυνοριακής αναγνώρισης και εκτέλεσης σε μέτρων προστασίας για αστικές υποθέσεις. Τώρα, ποιο είναι το νομικό αγαθό που είναι αντικείμενο προστασίας. Είναι η ελευθερία, είναι η ψυχική και σωματική ακεραιότητα Τώρα αυτά τα αγαθά, από τη στιγμή που αυτά τα αγαθά ε, βρίσκονται σε κίνδυνο, θα προσπαθήσουμε να τα προστατεύσουμε με την πρόταση αυτή του κανονισμού. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που διέπει και τους άλλους κανονισμού, είναι ο περιορισμός των λόγων για άρνηση. Αν έχουμε ένα πιστοποιητικό που θα γίνεται κοινώς αποδεκτό, δεν θα μπορεί ένα κράτος που καλείται να εκτελέσει αυτό το πιστοποιητικό να αρνηθεί την εφαρμογή, την εκτέλεση. Μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις αντιφατικών αποφάσεων και μάλιστα σε καταστάσεις που είναι σαφώς οριοθετημένες στην πρόταση, μπορούμε να δεχτούμε την πιθανότητα άρνησης εκτέλεσης του μέτρου προστασίας. Κάτι άλλο σημαντικό εδώ, μια και μιλούμε για ταχύτητα και πόσο σημαντικό είναι ο χρόνο, είναι το θέμα τη ε, κατάργηση του περιορισμού των διατυπώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να μην ε, ζητούμε επιπλέον διατυπώσεις σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας. Γιατί το δίκαιο ε, το εφαρμοστείο δίκαιο φυσικά θα είναι το δίκαιο ε, που γνωρίζουν οι δικαστές, οι ανακριτές. Είναι το δίκαιο του κράτους που εφαρμόζει αυτό την, ε, τη λύση και νομίζω ότι η πρόταση αυτή για το εφαρμοστείο δίκαιο είναι πολύ καλή. Και κάτι άλλο που το μεταλαμπαδεύσαμε από την ε, λογική της Δικαστική συνεργασία στι αστικέ υποθέσει είναι η χρήση των τυποποιημένων εγγράφων. Είναι σημαντικά τα τυποποιημένα εγγράφα για να εξασφαλίσουν ταχύτητα, ομοιομορφία και να επιλύσουν και κάποια γλωσσικά προβλήματα που είχαμε στον τομέα αυτό. Η χρήση τυποποιημένων εγγράφων είναι θεμελιώδης σημασία. Στην δική μου μελέτη αναφέρω και κάποιες επικρίσεις των λύσω, κάποιες κριτικές. Πάντως η γενική ιδέα, η κεντρική ιδέα είναι ε, καλή και δεν θέλω να σας, να σπηλώσω αυτή τη θελκτικότητα της πρότασης, να μην χαλάσω το σεξ χαρακτήρα της. Ευχαριστώ. Έχω δει ότι υπάρχουν διάφοροι που θέλουν το λόγο, αλλά θα συζητήσουμε στο τέλος του τμήματος αυτού της διαδικασίας. Οπότε να δώσω τώρα το λόγο για τις, ε, στον ομιλητή για τις διασυνοριακές επιπτώσεις ε, της νομικής προστασίας των ενηλίκων. Οπότε δεν ξέρω να δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Δυστυχώς φεύγει το αεροπλάνο μου. Θα ήθελα να πω κάτι πολύ σύντομα. Πολύ γρήγορα παρακαλώ. Είμαι η Άννα Χόλμ, είμαι Φιλανδή ε, βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να κάνουμε βήματα για να βελτιώσουμε την ε, προστασία των θυμάτων. Όταν μιλάμε για τις διαταγές προστασίας ή απομάκρυνσης, που, που πρέπει να αναγνωρίζονται και σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να το αναγνωρίζουν τα άλλα ε, κράτη. Ε, ε, γιατί όπως ξέρετε στη Φιλανδία τέτοιες εντολές διαταγές απομάκρυνσης δεν μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς να υπάρχει κάποια καταδίκη. Με αυτό το νέο όργανο που έχουμε τώρα είναι δυνατόν να καλύψουμε, να συμπεριλάβουμε και αυτές τις διαταγές απομάκρυνσης. Η Φιλανδία περιμένει, θα ήθελε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και σε ένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη χρήση αυτού του μέσου. Ένα άτομο που μπορεί να είναι επικίνδυνο για άλλους δεν ε, γνωρίζω ορισμένε φορές για ποιε χώρε ισχύει κάποια εντολή απομάκρυνσης. Στόχος μια τέτοια εντολή είναι να μην υπάρξει βία κατά του θύματος. Οπότε είναι βασικό το άτομο που είναι υποκείμενο μιας τέτοιας διαταγή να ξέρει σε ποιες χώρε ισχύει, ποιε χώρε το αποδέχονται. Να ξέρει λοιπόν σε ποιε χώρε δεν μπορεί να πάει. Οπότε ζητήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση να εμβαθυνθεί η μελέτη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Για το επόμενο θέμα τώρα, για την ε, νομική προστασία των ενηλίκων, έχουμε δύο που θέλουν να πάρουν τον λόγο για τη διάσκεψη της Χάγης. Είστε από τη διάσκεψη της Χάγης, θα μιλήσετε και οι δύο. Μισή παρακαλώ λοιπόν παρέμβαση ο καθένας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προβουλευτές, κύριοι εμπειρογνώμονες, ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σε αυτό το σεμινάριο. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα. Πάντα αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία συνεργασία. Ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα. Πρώτον, η σύμβαση της Χάγης ε, του 2000 και οι συνάδελφοι θα πούν κάτι μετά για τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2006 για τους ενήλικες. Αν δείτε έξω, δεν μπορεί παρά να σκεφτείτε πόσο σκόπιμο είναι να μιλήσουμε τώρα, πόσο επίκαιρο είναι να μιλούμε για την προστασία των ενηλίκων. Τι σχέση έχει αυτό με τον καιρό, θα αναρωτηθείτε. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο οι χειμώνες είναι και πιο κρύοι. Υπάρχει πολύ σπάγος στα πεζοδρόμια. Οπότε είναι επικίνδυνα τα πεζοδρόμια για τους ηλικιωμένους. Οπότε οι πιο εύποροι ηλικιωμένοι πάνε στις νότιες χώρες μετακομίζουν εντός της Ευρώπης αλλά και εκτός όπως είδαμε και όπως μας λένε οι, οι δήμονες για την ε, κλιματική αλλαγή πηγαίνουν ε, στην Τινησία, το Μαρόκο και ε, υπάρχει ένα διεθνές μέσο για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό διότι όσο μεγαλώνουμε μπορεί να αποκτήσουμε κάποια αναπηρία. Και αν συμβεί αυτό, πρέπει να γνωρίζετε ποιος έχει δικαιοδοσία, ποιος νόμος θα εφαρμοστεί και πώς οι αποφάσεις θα αποφασιστούν, οι αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος να έχει την επιμέλειά σας κάποιος να αναλάβει τη φροντίδα για τις ε, προσωπικές σας ανάγκες και τα περιουσιακά σας στοιχεία κινητά και ακίνητα. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που θα βοηθήσουν την επίλυση των θεμάτων αυτών. Ο επόμενος εμπειρογνώμων, κύριος Φρίμστον, βεβαίως θα εξηγήσει ότι ναι δεν είναι τέλεια η σύμβαση γιατί δεν ορίζονται κάποιοι όροι εμείς απαντάμε ότι αυτή η έλλειψη ακρίβειας ε, στην πραγματικότητα είναι προτέρημα, γιατί για να καταλήξουμε για το τι είναι ε, αναπηρία, τι είναι ανεπαρκή μέσα κτλ. είναι δύσκολο μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου. Το βασικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη οι δικαστές να μπορούν να εξετάζουν τις καταστάσεις με βάση το εθνικό τους δίκαιο και να λαμβάνουν αποφάσεις ότι αυτό είναι αναπηρία, αυτό είναι δυσχέρεια. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις αποφάσεις τους. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη λήψη μέτρων προστασίας από ένα κράτος που να αναγνωρίζονται και να εκτελούνται και σε άλλα κράτη-μέλη. Βεβαίως υπάρχουν όλες οι αναγκαίες διαδικαστικές εγγυήσεις ούτω ώστε να υπάρχει σωστή αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων. Έξι χώρες μέλη υπογράφουν αυτή τη συμφωνία, Τσεχία, Εστονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο για τη Σκοτία. Και 7 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση, Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Πολωνία. Το 2008 υιοθετήθηκε ένα πόρισμα του Συμβουλίου που συνιστούσε οι χώρε που έχουν υπογράψει να επικυρώσουν όσο να το πιο σύντομα αυτή τη σύμβαση και όσοι δεν έχουν υπογράψει να υπογράψουν το συντομότερο. Ένα αντίγραφο αυτή τη απόφαση του Συμβουλίου έχει διανεμηθεί στου ευρωβουλευτέ και του εμπειρογνώμονε. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση. Υπάρχει ανάγκη κανόνων στον τομέα αυτό και εντό τη Ένωση αλλά και διεθνώς. Γιατί όπως είπα, οι πιο εύποροι ηλικιωμένοι πηγαίνουν σε θερμότερα κλίματα. Πιο ευχάριστα. Καταληκτικός πώς. Κάτι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Αν θα είχατε το, τη δυνατότητα να εγκρίνετε μια ευρωπαϊκή εξουσία ε, νομικού αντιπροσώπου, να έχουμε δηλαδή χώρο, ξέρετε αυτό, αυτή η δυνατότητα power of attorney είναι μια ε, δυνατότητα που δίνει το common law της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά υπάρχουν παρόμοιες ε, ρυθμίσεις στην ε, Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και στην Ελβετία. Δυνατότητα εκπροσώπησης μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ούτω ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή της σύμβασης. Επειδή ε, ξέρω ότι πολλά άτομα από το Καναδά πάνε στην Αριζόνα ε, γιατί είναι πολύ ε, πιο καλό το κλίμα εκεί. Ξέρω ότι αυτά τα άτομα έχουν ανάγκη εκπροσώπηση και προστασία. Σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα γιατί τον καθυστέρηση. Ναι, βεβαίω, ε, πολύ σύντομα για την ε, σύμβαση του 2006 των ΗΠΑ για τα άτομα με αναπηρία και την ε, Σύμβαση 2000 της Χάγης η πιο πρόσφατη. Είναι η πιο πρόσφατη λοιπόν ε, η σύμβαση αυτή των Εθνών. Ο στόχος της ε, σύμβασης αυτής είναι να προωθήσει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει την πλήρη δυνατότητα όλα τα άτομα με αναπηρία να απολαμβάνουν πλήρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να γίνεται σεβαστή η αξιοπρέπειά τους. Από τότε που εθετήθηκε αυτή η σύμβαση έχει προκαλέσει 155 υπογραφές και 120 χώρες μέλη παγκόσμια την έχουν υιοθετήσει. Όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν υπογράψει αυτή τη σύμβαση και 24 κράτη την έχουν ήδη επικυρώσει. Η σύμβαση Χάγη 2000 είναι μια πολύτιμη ευκαιρία για τα κράτη που είναι μέλη του, της Σύμβασης του 2006 να εφαρμόσουν τις ευρύτερες υποχρεώσεις που απορρέουν από την ε, Σύμβαση του 2006 για τα άτομα ακριβώς με αναπηρίες που είναι υποκείμενο της Σύμβασης του 2000. Αυτή είναι τώρα η γενική περιγραφή που έχετε ήδη λάβει τη Σύμβαση του 2000 που παρέχει περισσότερη προστασία και ε, νομική ασφάλεια για ε, άτομα που είναι ευάλωτα με βάση τους ορισμούς. Και βεβαίως οι δύο συμβάσεις πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως για παράδειγμα διατάξεις του άρθρου 18 για την ελεύθερη διακίνηση, ελεύθερη ηθαγένεια, το άρθρο 32 για διεθνή συνεργασία, το 12 για την ε, ίση αναγνώριση και ισότιμη μεταχείριση έναντι του νόμου Επίσης ε, άρθρα για την αξιοπρέπεια των ατόμων αναπηρία, το 25 για την υγεία, 13 πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οπότε, καλούμε τα κράτη-μέλη της Ένωσης να εξετάσουν ε, πώς μπορούν να ε, δουλέψουν από κοινού αυτά τα δύο σημαντικά διεθνή μέσα, ούτω ώστε να υπάρξει ευρεία επικύρωση της Σύμβασης Χάγη 2000. Σας ευχαριστώ που αυτό το σύντομα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φρίνστον. Ευχαριστώ. Σας παρακαλούσα μάλλον να παρουσιάσετε ποιον εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας είμαι ευγνώμων που με καλέσατε. Σύντομα θα ήθελα να φεδώ στην πρακτική εμπειρία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί να καταλήξω στα συμπεράσματά μου. Είναι περίπλοκο το θέμα της ε, ικανότητας αναπηρίας. Δεν είναι κάποια ξεχωριστή νομική ταξινόμηση διότι για διάφορα επίπεδα, για διάφορες πράξεις απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. Για να υπάρχει ας πούμε το δίκαιο για τη σύναψη συμβάσεων, κανονισμός για την διαδοχή, για την κληρονομιά, η δυνατότητα να είναι κανείς ικανός να συντάξει μια διαθήκη εξαρτάται από το αν θεωρείται ικανός. Λοιπόν, η σύμβαση της Χάγης είναι πραγματικά μια υπέροχη προσθήκη ε, στο ιδιωτικό δίκαιο, διεθνές ιδιωτικό δίκαιο και ασχολείται με μέτρα προστασίας, οπότε εφαρμόζει τους κανόνες περί δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου και ε, αναγνώρισης και εφαρμογής που εφαρμόζονται στα μέτρα προστασίας. Επιπλέον, καθορίζονται κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τη δυνατότητα εκπροσώπησης για την εξουσιοδότηση μέσω δικηγόρου. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Σκοτία επικύρωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο επικύρωσε την ε, σύμβαση για την Σκοτία αλλά όχι για την Ουαλία και την Αγγλία. Εσωτερικά έχουμε την ίδια νομοθεσία και είχαμε κάποιες υποθέσεις στις οποίες εξετάστηκε ποια επίπτωση είναι της σύμβασης και είναι πάρα πολύ επικοδομητικό αυτό. Ίσως θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Φιλίπ. Δηλαδή θα ήθελα να πω ότι η Σύμβαση της Χάγης ως προαναφέρθηκε σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε αυτό το τομέα νομίζω ότι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός είναι κάτι που απαιτείται δηλαδή η δυνατότητα νομικής εκπροσώπησης, εξουσιοδότησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζεται αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο όπως αναφέρθηκε σε με μέσα δεν υπάρχει η αναγνώριση της εξουσιοδότησης μπορεί να έχει την αποδοχή αυτής της εξουσιοδότησης τι σημαίνει αποδοχή, η λέξη αποδοχή ε, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα στην Ευρώπη όσον αφορά την εξουσιοδότηση τη νομική μέσω δικηγόρου. Δείχνουν τα προβλήματα ότι στην αρμόδια, το να αποδείξει ότι ισχύει αυτή η έγκριση, αυτή η εξουσοδότηση στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστεί. Γι' αυτό παροτρύνω την Επιτροπή και τα Εθνικά Κοινοβούλια και σας λέω παρακαλώ, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη θα επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση, διότι είναι χρησιμότατη. Θα έλεγα σχεδόν σεξι. Αλλά πέραν αυτού, θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον δεχόμενο κανονισμό και να εξετάσει την ιδέα ευρωπαϊκής εξουσιοδότησης νομικής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους ενήλικες ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Τελευταία παρέμβαση όσον αφορά αυτό το θέμα, ο ε, κύριος Φιωρίνη, για τη νομική βάση για το οικογενειακό δίκαιο. Ποια νομική βάση για το οικογενειακό δίκαιο είναι το θέμα. Έχετε ένα δεκάλεπτο περίπου και μετά συζητήσουμε, κυρία Φιωρίνη. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε αυτό το δεκάλεπτο που μου δίνετε. Πριν ε, ε, αρχίσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Νομική Επιτροπή για την οργάνωση της ημερίδας αυτής της μελέτης. Η εξέλιξη στο οικογενειακό δίκαιο, συνεχίζω στα αγγλικά, ήταν εντυπωσιακέ. Το 2000, για παράδειγμα, είχαμε μόνο την εφαρμογή της ε, Σύμβασης των Βρυξελών για τις υποχρεώσεις ε, ε, διατροφής. Ενώ σήμερα έχουμε ένα ευρύο πλωστάσιο διατάξεων οικογενειακού δικαίου και μάλιστα αναμένεται να εγκριθούν πολύ περισσότερες. Και όπως ακούσαμε και προηγουμένως, υπάρχουν περιπτώσεις διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου που καλύπτονται από εθνικούς κανόνες. Αν λοιπόν θέλουμε να ολοκληρώσουμε το χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης, ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική βάση για τις πρωτοβουλίες ε, που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο βασικούς κανόνες με διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι στο παρελθόν. Καταρχήν, είναι δυνατόν να, χρησιμο... να θεσπιστούν πανευρωπαϊκά μέτρα με βάση το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί σε επίπεδο οικογενειακού δικαίου ισχύει μια ειδική νομοθετική διαδικασία. Απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο και μάλιστα προηγούμενη διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, είχαμε τη ρήτρα Πασαρέλα για την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Δεύτερη διάβλος είναι η λήψη μέτρων που δεν θα καλύπτουν το σύνολο της ε, επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα, ε, ισχύσουν, θα ισχύσουν μόνο οι ορισμένες χώρες μέλη. Για παράδειγμα, ενισχυμένη συνεργασία, για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ συγκεκριμένου αριθμού κρατών μελών. Και στην περίπτωση του οικογενειακού δικαίου Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την ειδική νομοθετική διαδικασία. Παρόλο που και πάλι χρειαζόμαστε μια ρήτρα γέφυρα, μια μεταβατική ρήτρα δηλαδή, όπως ε, η ρήτρα Πασαρέλ που ανέφερα προηγουμένως, που χρήζει όμως διαφορετικής νομικής βάσης. Υπάρχουν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις λοιπόν. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το άρθρο 81, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο και την ειδική νομοθετική διαδικασία. Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει με εξαιρέσει τη διαδικασία, ότι η διαδικασία απόφαση δεν ε, ισχύει για οικογενειακά θέματα, για θέματα οικογενειακού δικαίου. Οπότε η ειδική μεταχείριση του οικογενειακού δικαίου εξαρτάται ή εξηγείται από την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει αυτό το θέμα και την ισχύ των εθνικών παραδόσεων ε, στο θέμα αυτό. Πάντως με και το θέμα της διαδικασίας διαβούλευσης μπορεί να αμφισβητηθεί για πολλά θέματα. Μάλιστα, σε ένα τομέα που είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, δεν θα πρέπει οι πρόσωποι τους να εμπλέκονται πιο ενεργά στη διαδικασία. Δεύτερον, η απέτηση της ομοφωνίας στο Συμβούλιο μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη, την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου η δυνατότητα ανησυχηρίας ε, χωρομελών και μια ψηφίες που μπορεί να μπλοκάρει ε, για λόγους εθνικού συμφέροντος τέτοιες πολιτικές. Είδαμε και στα πλαίσια του κανονισμού Ρώμη 3 παρόμοιες συμπεριφορές. Τώρα, κάποιοι συμβασμοί που δεν είναι ικανοποιητικοί μπορεί να αλλοιώσουν και να εξουδετερώσουν μια πολιτική υπέρ της οικογένειας. Και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 μπορεί ε, να ε, αμφισβητεί τη δυνατότητα της ε, θέσπισης παρευρωπαϊκού δικαίου ή της υλοποίησης των στόχων. Πάντως, η χρήση της ρήτας πασαρέλας θα πρέπει να προωθηθεί ως εναλλακτική λύση. Με βάση το άρθρο 81, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, το Συμβούλιο μπορεί ομόφωνα και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει ότι κάποιε πτυχέ του οικογενειακού δικαίου διασυνοριακή εφαρμογή μπορεί να θεσπιστούν με την συνήθη νομοθετική διαδικασία, κάτι που προποθέτει μεγαλύτερο διοργανικό διάλογο, πιο εντατικό και ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, όχι ομοφωνία. Οπότε θα μπορούσε να διαρωτηθεί κανεί τα αποτελέσματα αυτά. Ε, για ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως είναι το οικογενειακό δίκαιο που επηρεάζεται από τις, ε, παραδόσεις, τις εθνικές παραδόσεις δεν θα πρέπει να ε, ακυρωθεί ε, εις βάρος της δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει οικογενειακό δίκαιο. Η Πασαρέλα αποδυναμώνοντας την κυριαρχία των κρατών μελών είναι επιχείρημα που δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά. Η Πασαρέλα του 81-3 απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο και έγκριση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οποιοδήποτε Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει βέτο στη χρήση αυτή τη διαδικασία. Οπότε, αν ένα προτινόμενο μέτρο θεωρηθεί ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και απειλεί ευαίσθητη εθνική πολιτική, η χώρα μέλος μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή της Ρήτας Πασαρέλας ε, είτε με το βέτο στο Συμβούλιο, είτε με την ε, απόρριψη από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Αν δεχτούμε τώρα επί της αρχής τη Ρήτρα Πασαρέλα, δεν είναι σίγουρο ότι οι υπόλοιπε ε, ε, οι υπόλοιπε πτυχέ του οικογενειακού δικαίου θα εμπέσουν στη συνήθεια διαδικασία. Τώρα, η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν αφορά τόσο το οικογενειακό δίκαιο όσο το περιεχόμενο του προτινόμενου μέτρου. Φαίνεται ότι σε πολλούς ε, τομείς υπάρχουν ε, στοιχεία του οικογενειακού δικαίου και στοιχεία του ενοχικού δικαίου ή στοιχεία του δικαίου για τη, της Οπότε ένας τομέας που δεν είναι μόνο αμυγός οικογενειακού τομέα δεν δικαιολογεί από μόνο του τη ρήτρα γέφυρα, τη ρήτρα πασαρέλα. Γιατί το ότι ένα τομέα είναι μεικτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο ευαίσθητο από ότι ένα αμυγή ε, τομέα του οικογενειακού δικαίου. Οπότε η σκοπιμότητα της χρήση της ρήτρα πασαρέλας και η ομόφωνη αποδοχή της εξαρτάται από το περιεχόμενο του προτινόμενου μέτρου η ρήτρα αυτή μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλη ανάλογα με το κατά πόσο ένα τομέα είναι ήδη έστω και μερικώ εναρμονισμένο, μέσω τη νομολογία του ΔΕΚ, για παράδειγμα, όπω ακούσαμε το πρωί, ή μέσω ε, κάποιων διεθνών νομικών συμφωνιών. Η χρήση της συνήθως νομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει να διευκολυνθεί και σε περιπτώσεις όπου το προτινόμενο μέτρο ε, ρητά ή έμεσα ή επί της αρχής έχει γίνει δεκτό ή είναι πιθανό να γίνει δεκτό από όλα τα κράτη-μέλη. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα. Οπότε ερχόμαστε στο επόμενο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα πανευρωπαϊκών μέτρων με την προώθηση της διαδικασίας της ενισχυμένης συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη περιλαμβάνει κάποιες ε, διατάξεις για την ενισχυμένη συνεργασία που συνοδεύονται όμως από πολλές προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να ε, εφαρμοστεί η ενισχυμένη συνεργασία. Βέβαια, ακόμη και να συντρέχουν οι προποθέσει, δεν είναι αυτόματη η εφαρμογή τη ενισχυμένη συνεργασία. Για να ενεργοποιηθεί η ενισχυμένη συνεργασία, απαιτείται πρόταση ε, που θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέτοιου είδους ενεργοποίηση της ενισχυμένης συνεργασίας ε, θα πρέπει να γίνει μόνο μετά από δελεχή εξέταση δύο πτυχών. Η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει πραγματικά να είναι το ίστατο μέτρο, η έσχατη λύση, πρώτον, και δεύτερον θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις δυσκολίες είναι ότι οι συνθήκες δεν καθορίζουν τι θα πει η έσχατη λύση. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, ο στόχος ενός μέτρου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλές πολιτικές εναλλακτικές εξίσου κατάλληλες. Για παράδειγμα, μία πρώτη τέτοια επιλογή, πολύ φιλόδοξη, θα ήταν η εναρμόνιση. Άλλη επιλογή πολιτικής θα ήταν μια πιο συντηρητική εκδοχή της ε, και οι δυο όμως βαίνουν στην υλοποίηση του ίδιου στόχου. Αν το προτινόμενο μέτρο επιλέξει την πρώτη επιλογή, και αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί ένα μέτρο ενισχυμένης συνεργασίας ε, για μέτρο της, πολιτικής, ε, της πρώτης πολιτικής επιλογής ε, να εφαρμοστεί. Να θεωρηθεί λοιπόν η λύση για την πραγματοποίηση του στόχου ή μήπως θα πρέπει να αναζητηθεί εναλλακτική λύση με βάση τη δεύτερη πολιτική. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, όλα αυτοί οι προβληματισμοί ε, εκφράζουν τις ανησυχίες για την ενισχυμένη συνεργασία. Το θέμα είναι, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε κανόνες που μπορούν να έχουν αποτέλεσμα περισσότερα, κάτι περισσότερο με τη χρήση λιγότερων, ε, λιγότερο υποχρεωτικών κανόνων ή το αντίθετο. Κυρία μου, θα πρέπει να ολοκληρώσετε κάποια στιγμή. Έχετε μακρηγορήσει. Καλώς, να ολοκληρώσω. Je... Θα ήθελα λοιπόν να, να καταλήξω σε δύο θέματα. Πολύ εύκολα ξεχνούμε ότι ε, στα πλαίσια του άρθρου 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται δύο διαφορετικοί στόχοι. Η στόχη ενός μέτρου και η στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στόχη ενός μέτρου ε, πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο και το δεύτερο καταληκτικό σχόλιο είναι ότι η επανειλημμένη χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας δύσκολο δικαιολογείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού, ενός ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου και δεν μιλώ για τις αρχές του, αλλά για τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενισχυμένη συνεργασία. Και ε, μια πληθώρα προσεγγίσεων ίσως δημιουργήσει έλλειψη ασφάλειας δικαίου και μια βεβαιότητα. Παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια δικαίου είναι προϋπόθεση ε, για την πραγματική απονομή της δικαιοσύνης. Οπότε η πολλαπλή εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας θα αποβεί εις βάρος ε, θεμελιώδου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι κατά τη γνώμη μου η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να εξεταστεί μόνο υπό εξαιρετικές περιστάσεις. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Έχουμε χρόνο για συζήτηση. Αν θέλετε θα σας δώσω το λόγο, αν ζητήσετε, να σας επισημάνω ότι έχουμε 25 λεπτά καθυστέρηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμά μας και υποθέτω ότι ίσως είχετε τρένα, αεροπλάνα να προλάβετε. Μπορείτε να πάρετε το λόγο όμως, ε? Non, personne, madame, vous Θέλατε εσείς να μιλήσετε κυρία μου ή όχι. Ορίστε, σας δίνω το λόγο. Κυρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Σύμβαση για την Προστασία των ελλήνων είναι η λογική συνέχεια της Συμβάσεως του 1996 για την Προστασία των Παιδιών. Η προστασία των παιδιών α, τελειώνει στα 18 και των ενηλίκων η προστασία ξεκινά από τα 18. Και αυτό που σημαντικό είναι να δούμε ότι τα κείμενα είναι πάρα πολύ παρόμοια. Οι δύο συμφάσει λειτουργούν παρομοίω για την επίτευξη των δύο στόχων. Αρκετέ χώρε τα τελευταία χρόνια επί μακρόν προσπάθησαν να εφαρμόσουν ε, τη σύμβαση του 1996. Ε, τα ενθαρρύνουμε να περάσουν και στην εφαρμογή της συμβάσεω του 2000. Ε, το έργο του προβληματισμού ήδη έχει γίνει, η ανάλυση και μπορούν να κερδίσουν πάρα πολύ χρόνο περνώντας στην εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για αυτή την ε, διευκρίνηση που είναι σημαντική. Θα παραχωρήσω την Προεδρία στην κυρία Κατρίν Τζαπόνε, η οποία θα προεδρεύσει σε αυτό το τελευταίο τμήμα. Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφε, που καθυστερημένα σας παραδίδω την Προεδρία σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, ίσως να είσαστε πιο αυστηροί από μένα όσον αφορά την, ε, τις παρεμβάσεις και τον χρόνο που παίρνουν. Um, Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο τμήμα του εργαστηρίου μας για το αστικό δίκαιο και δικαιοσύνη. Διαρευνούμε το θέμα του κατά πόσο οι Ευρωπαίκες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απολαμβάνουν ε, ελεύθερη, ελεύθερη μετακίνηση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και μετά θα συνεχίσω με την ε, Προεδρία και θα ακολουθήσουμε τη σειρά με τους τελευταίους ομιλητές που έχουν προγραμματιστεί. Είναι το τελευταίο τμήμα μιας πολύ μακράς ημέρας, αλλά παρακαλώ να προσέξετε, να ακούσετε και να αποφεληθείτε από τα όσα μας πούν οι εμπειρογνώμονές μας, που θα μιλήσουν σε λίγο. Λοιπόν, κάποια αναρκτήρια σχόλια. Ε, το θέμα ε, της οικογενειακής καταστάσεως συνδέεται πολλές φορές με το θέμα της ταυτότητας, με τα πολιτικά δικαιώματα, το σχετικό κανονισμό και την ε, αναγνώριση του ατόμου από το κράτος και την κοινωνία γενικότερα. Το θέτο ότι μια τέτοια αναγνώριση θυγραμμίζεται είναι αποτέλεσμα πολιτισμικών προδιαγραφών ή παραδοσιακών πρακτικών. Αλλαγή σε αυτόν τον τομέα της νομοθεσίας μπορεί να είναι αργή, όμως αλλαγή στην μορφή διασυνοριακής διαβίωσης και εργασίας είναι κάτι που προχώρησε αρκετά γρήγορα όπως γνωρίζουμε μετά την αρχή της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Η πραγματικότητα είναι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν διάφορους κανόνες περί οικογενειακής καταστάσεως στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν η αναγνώριση της οικογενειακής κατάστασης ε, παρεμποδίζεται είναι πάρα πολύ επαχθής Όπω είδαμε και από προηγούμενε παρεμβάσει, οι πολίτε Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρω ε, το δικαίωμα ελεύθερη μετακίνηση και αυτοί οι περιορισμοί επί του πολίτου μπορούν να έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσμα, ε, συνέπεια όσον αφορά την ταυτότητά τους, την οικογένειά τους, την απασχόλησή τους. Τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να εξισορροπούνται με την ανάγκη ε, της καταπολέμησης της απάτης όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα μας από το θέμα. Στην Ιρλανδία, παραγματος χάρη, η νομοθεσία ε, ετοιμάζει το νομοσχέδιο για να αντιμετωπίζει τους συμβατικούς γάμους. Μετά από ανησυχίες που εξεφράστησαν για ε, γάμους με πολίτες, ε, με υπηκούς, αυτού του τύπου γάμους, υπηκούς άλλων χωρίς Ευρωπαϊκής Ενώσεων, τη Ενώσεω και τρίτε χώρε. 350.000 γάμοι γίνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα επηρεάζονται πολύ από, αυτό, από αυτού του γάμου. Και προσωπικά θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Είμαι Ιρλανδέζα επίκος και έχω και την υπηκότητα των ΗΠΑ. Διαμένω στο Δουβλίνο με τον σύζυγό μου, ε, δόκτωρ και ε, κυρία Λουίς Γκίνιγκαν και προσπαθώ να αναγνωριστεί ο πολιτικός μου γάμος ε, με τον Δόκτωρα Γκίλιγκαν στην Ιρλανδία. Είναι καναδικός γάμος και παντρευτήκαμε στον Καναδά πριν από 8 χρόνια. Ήταν το μόνο μέρος στον κόσμο που θα μπορούσα να παντρευτώ με την σύζυγό μου τότε, χωρίς να είμαστε υπήκοοι εκεί. Αντιμετωπίσαμε παρόμοιες ε, ε, δυσκολίες με άλλα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, με άλλους πολίτες Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής αν φύγουν τη δικαιοδοσία στην οποία ανέλαβε χώρα ο γάμος τους. Στην Ιρλανδία η πολιτική γάμη ομοφιλοφίλων ζευγάρων από εδώ, από το Βέλγιο ή από οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που προβλέπει ισότητα, ισότιμη αναγνώριση θα μετατραπόταν στην Ιρλανδία σε νόμιμη συμβίωση που δίνει λιγότερα δικαιώματα από ότι ένας βελγικός γάμος και θα θεωρούσε ότι τότε αυτή η μετακίνηση οδηγεί σε υποβάθμιση της οικογενικής καταστάσεως. Τα οικογενειακά αυτά, η οικογενική κατάσταση αφορούν τον πυρήνα της ταυτότητας. Σάγια αρουσιαστής και νομοθέτη στην Ιρλανδία πολύ συχνά το ανέφερα αυτό για την αναγνώριση του φίλου για άτομα φιλομεταβατικά. Η Ιρλανδία είναι μία από τις μόνες αναπομένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν αναγνωρίζει ε, το φύλο των φιλομεταβατικών. Ενώ άτομα αυτής της κατηγορίας αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα και οι του. τους. Πάνω από 12 εκατομμύρια άτομα ζουν και μελετούν σε αυτή τη χώρα και δεν είναι ε, ε, υπήκοοι της χώρας. Όσοι έχει το κοινοτικό δίκαιο σε αυτή τη φάση, η οικογενειακή κατάσταση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, όταν τα κράτη-μέλη εξασκούν αυτή την αρμοδιότητα πρέπει να συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τι διατάξει τη συνθήκη για την ελευθερία που έχει κάθε πολίτη τη Ένωση να μετακινείται και να διαμένει ε, στην επικράτεια των κρατών μελών. Για το τελευταίο αυτό τμήμα λοιπόν συζητήσεις θα εξετάσουμε ποια είναι τα παρόντα εμπόδια που υπάρχουν και το δεχόμενο μέλλον για την οικογενειακή κατάσταση, καταχώρηση οικογενειακή κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας βοηθήσει σε αυτό θα ακούσουμε, να μας βοηθήσουν, θα ακούσουμε τις εμπειρογνώμονες. Καταρχάς, η δόκτωρ Μαριολίνα Ελιαντώνιο που είναι σύμβουλος όσον αφορά μια εταιρεία ε, στη, που παρέχει νομικές συμβουλές στις Βρυξέλλες και θα μας μιλήσει για την οικογενική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι τα πιο κατεπήγοντα προβλήματα της πολίτης της Ευρωπαϊκής και την ανάγκη που υπάρχει για να γίνει κάτι, για να υπάρξει δράση. Και σας δίνω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Χαίρομαι που ξεκινήσατε ε, υπογραμμίζοντας το, την, είναι πολύ επίκαιρο το θέμα αυτό της οικογενειακής καταστάσεως ε, η πλειοψηφία πιστεύω των παρόντων στην αίθουσα ε, αντιμετωπίζει μια διασυνοριακή κατάσταση διότι το διασυνοριακό καθεστώς μπορεί να προκύπτει διότι κάτι από εμά ζούμε στο εξωτερικό παραδείγματο χάρη αποδείχθηκε το 2010 πάνω από 12 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος αλλά οι διασυνοριακές αυτές καταστάσεις δημιουργούνται διότι και κάποιος έρχεται στις Βρυξέλλες για μια διάσκεψη, για να επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο ή, ε, ή υπάρχουν καταστάσεις ευτυχής ή λιγότερο ευτυχής Παραδείγματο χάρη επίσκεψη σε, σε γιο ή κόρη που γεννά στο εξωτερικό ή γιατί πεθαίνει κάποιο στο εξωτερικό. Μπορεί να προκύψουν αυτέ τι καταστάσει. σω και για μια σύντομη διαμονή στο εξωτερικό, για εργασία. Έχουμε δει ότι πέντε από χίλιου εργαζομένου μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι διασυνοριακοί μετακινούμενοι εργαζόμενοι. Αντιμετωπίζουν καθημερινά μια διασυνοριακή κατάσταση ή ε, μπορεί να είναι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που αντιμετωπίζουν οι συνοριακέ καταστάσει για λόγου ε, τουρισμού. Το 2010, παραδείγματο χάρη, πάνω από 90 εκατομμύρια πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση επισκέφτηκαν άλλο κράτο μέλο για τουρισμό ή για την παροχή, για τη λήψη υπηρεσία, να πάνε για περίθαλψη σε νοσοκομείο, στον οδοντογιατρό. Υπάρχει ποικιλία καταστάσεων διασυνοριακού χαρακτήρα που μπορεί να προκύπτουν για την καθημερινή ζωή του καθεμιανού και σε κάθε μια τέτοια μετακίνηση διασυνοριακή οι πολίτες, ο καθένας από εμά ίσως να χρησιμοποιηθούν έγγραφα που πιστοποιούν την οικογενειακή του κατάσταση, πιστοποιητικό γέννηση, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό θανάτου. Ε, όλα αυτά είναι βασικά έγγραφα που ο καθένας από εμά πρέπει να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικά για να έχει κανείς πρόσβαση σε πολλές άλλες υπηρεσίες. Παραδείγματο χάρη να έχει κανείς πρόσβαση στο επίδομα ενεργείας Σε κάθε τέτοια διασυνοριακή περίπτωση, κατάσταση, οι πολίτες όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν θέματα που ζητούν, απαιτούν έγγραφα οικογενικής καταστάσεων, που αντιμετωπίσουν προβλήματα και εμπόδια. Γι' αυτό λάβαμε σαν μιλίο, σαν συμβουλευτικό φορέα, αναλάβαμε το καθήκον, μα το ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσουμε ε, τα, ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζονται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα οικογενειακής καταστάσεως σε διασυνοριακό πλαίσιο. Γι' αυτό διενεργήσαμε μία επισκόπηση ε, της νομολογίας της Ευρωπαϊκής και της γενικότερης για θέματα αστικού δικαίου και κάναμε συγκριτική μελέτη των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών και νομολογίας κάποιων επιλεγμένων ε, κρατών μελών. Επ' αυτής της βάσης εντοπίσαμε κάποια από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση σε διασυνοριακά πλαίσια και προσπαθήσαμε να προτείνουμε κάποια πράγματα, να κάνουμε κάποιες συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που να εμπίπτουν οι συστάσεις αυτές της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα βασικά αποτελέσματα, τα πορίσματα της μελέτης. Το πρώτο πρόβλημα που διαπιστώσαμε, πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας από εμά σε διασυνοριακές περιστάσεις είναι να καθορίσουμε πού, πού ακριβώς βρίσκονται τα έγγραφα αυτά της οικογενειακής κατάστασης. Ας πούμε ότι είμαι Ιταλίδα και πρέπει για οποιοδήποτε σκοπό να βρω το πιστοποιητικό γέννησης του πατέρα μου που γεννήθηκε στη Γερμανία. Το θέμα είναι το πιστοποιητικό γέννησης βρίσκεται εκεί που γεννήθηκε ο πατέρας μου ή εκεί που έζησε ο πατέρας μου για το υπόλοιπο της ζωής του ή εκεί που πέθανε. Α φανταστούμε ότι είναι τρει διαφορετικές πόλεις στη Γερμανία. Ίσως να μην γνωρίζω, ε, διότι δεν ξέρω πώς καλύπτει η Γερμανία το πώ διατηρούνται και φυλάσσονται τα διάφορα έγγραφα, πώς το αντιμετωπίζει. Κάθε κράτο μέλος βέβαια έχει δικούς του κανόνες σχετικά με την ε, φύλαξη αυτών των εγγράφων, αλλά για μένα που είμαι ξένη να πρέπει να βγάλω άκρη και να βρω που είναι το έγγραφο, ίσω να με μπερδεύει, να είναι κάτι χρονοβόρο και ίσω να είναι και κάτι δαπανηρό για μένα. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να μειώσει το βάρο των πολιτών. Καταρχάς θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν τους πολίτε περί των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κράτο μέλο για το πού φυλάσσονται τα έγγραφα. Υπάρχουν ιστοσελίδες όπως ε, της Ευρωπαϊκής για την νομική βοήθεια. Μπορεί να θαρρυνθούν τα κράτη-μέλη να έχουν σημεία επαφή σε εθνικό επίπεδο τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με το που φυλάσσονται έγγραφα. Μέσω ιστοσελίδας, μέσω νέας ιστοσελίδας, μέσω αριθμού τηλεφώνου κλπ. Α, ας φανταστούμε ότι έχω εντοπίσει τώρα εγώ που Υπάρχει ένα έγγραφο οικογενειακής κατάστασης. Πού φυλάσσεται. Το επόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ευρωπαίος πολίτης είναι το εξή. Αυτό το έγγραφο πώς θα κυκλοφορήσει. Πώς θα διανεμηθεί. Ας φανταστούμε το εξή. Εγώ και ο σύντροφο μου και οι δύο Ιταλοί θέλουμε να παντρευτούμε στις Βρυξέλλες. Και οι βελικές αρχές μα ζητούν πιστοποιητικό γέννησης για να μπορέσουμε να παντρευτούμε στο Βέλγιο. Ο μόνος τρόπος για να πάρω εγώ το Ιταλικό πιστοποιητικό γέννηση είναι να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στην Ιταλία, να πάω εκεί που φυλάσσεται το πιστοποιητικό γέννηση, να το πάρω, να επιστρέψω στο Βέλιο και να το υποβάλω στι βελγικέ αρχέ. Προφανώ αυτό είναι κάτι επαχθέ, δύσκολο, δαπανηρό για τον πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Η αδίποτε σύσταση περί του θέματος αυτού, δηλαδή πώς να μπορούν να ε, χορηγούνται με πιο εύκολο τρόπο και να κυκλοφορούν αυτά τα έγγραφα μεταξύ κρατών μελών έχει σαν στόχο τη μείωση του κόστους και τη μείωση του άχθους για τους πολίτες ενώ ταυτόχρονα, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, πρέπει να παραμένει το σύστημα αξιοπιστό και ασφαλές, το σύστημα με το οποίο κυκλοφορούν αυτά τα έγγραφα. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες ανταλλαγής ε, εγγράφων και αν αυτή τη ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολύνει τα κράτη-μέλη να τα διευκολύνει ε, στο να δημιουργήσουν αυτή την ηλεκτρονική βάση, την πλατφόρμα ή στο πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα υπάρχουσες πλατφόρμες. Ένα παράδειγμα από τις πλατφόρμες που υπάρχουν, ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την ε, διακίνηση τέτοιων ε, εγγράφων οικογενειακή κατάσταση υπάρχει. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο του Μητρώου για την Οικογενειακή Κατάσταση, το ICCS, ε, η Διεθνή Σύμβαση Υπαριθμών 33 για, το, για την οικογενειακή κατάσταση. Από τη στιγμή που θα έχω εντοπίσει τώρα εγώ που βρίσκεται το έγγραφο, μπορώ να το διανύμω, να το μεταβιβάσω και το επόμενο εμπόδιο είναι η επίσημη αναγνώριση ενός εγγράφου που αφορά την οικογενειακή κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό. Έχω πάρει εγώ το έγγραφό μου για την οικογενειακή μου κατάσταση, ας πούμε πιστοποιητικό θανάτου. Θα έχω ιταλικό πιστοποιητικό θανάτου που θα πρέπει να αναγνωριστεί στη Γερμανία, να θεωρηθεί ότι πράγματι είναι πιστοποιητικό θανάτου. Αν έτσι είχαν τα πράγματα, ένας Ιταλός πολίτης θα έπρεπε να μεταφράσει το έγγραφο στα γερμανικά από αναγνωρισμένο μεταφραστή, αναγνωρισμένο από τις γερμανικές αρχές. θα έπρεπε η σφράγιση και η έγκριση, η επικύρωση χρειάζεται στα διάφορα κράτη-μέλη του εγγράφου, αλλά είναι κάτι δαπανηρό και χρονοβόρο, διότι πολλές ε, αρχές εμπλέκονται, ε, χρειάζονται πολλές ανταλλαγές πληροφοριών, ε, πριν το έγγραφο αυτό να αναγνωριστεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα επικύρωσης, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια γενικότερη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω πάνω σε αυτό. Κατά πόσο και αν είναι δυνατόν να καταργηθεί αυτό το σύστημα, επικύρωση που απαιτείται, ίσως αργότερα θα μπορούσαμε να ακούσουμε στο πάνελ στη συζήτηση ποια είναι τα προβλήματα με τις απάτες που διαπιστώνονται. Η κατάργηση τώρα αυτού του συστήματος επικύρησης έχει έχει προταθεί από τη σύμβαση ICC υπαριθμών 17, κάτι που έχει ήδη κυρωθεί από αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γίνεται μια κίνηση προς την απλούστευση, ήδη έχει ξεκινήσει. Ταυτόχρονα όμως η σύμβαση των Βρυξελών είναι εφαρμοστέα σε έξι κράτη-μέλη όσον αφορά την κατάργηση του συστήματος επικύρωσης και υπάρχουν και διμερείς συμφωνίες. Άρα η ανάγκη περί απλουστεύσεως είναι ήδη αισθητή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολύνει ούτω ώστε να γίνει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς να πλουστευτούν ε, τα πράγματα. Εναλλακτική λύση να μην καταργηθεί αυτή η επισημείωση, να αντικατασταθεί ε, ε, αντί επί χάρτου να γίνεται ηλεκτρονικά αυτή η επισημείωση ηλεκτρονικό σύστημα υπάρχει, τέτοιο πρόγραμμα για επικύρωση και επισημείωση, το δημιούργησε η Σύμβαση τη χάγη για το Ιδιωτικό διεθνέ Δίκαιο και θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία ή παράδειγμα για αυτόν τον σκοπό. Εναλλακτικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δράσει σαν ε, φορέας διευκόλυνση για τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ούτω ώστε το σύστημα αυτό επισημείωση να γίνει αποτελεσματικότερο και λιγότερο χρονοβόρο και λιγότερο δαπανηρό και θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί πανευρωπαϊκή τεχνική λύση μέσω χρηματοδότησης, μέσω διευκόλυνσης της συζήτησης επ' αυτού του θέματος. Όσον αφορά τη μετάφραση, ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν ήδη υπάρχοντα πολύγλωσσα έντυπα. Η ICC έχει ήδη μια σύμβαση όσον αφορά τα πιστοποιητικά γάμου, γέννηση και θανάτου, να είναι πολύγλωσσα τα έντυπα και αυτό μπορεί να αποτελέσει την βάση για μια γενικότερη συζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για έντυπα τέτοια πολύγλωσσα. Θα μπορούσε μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα πρότυπο έντυπο πολύγλωσσο αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το, ε, το πιστοποιητικό γέννηση έχει την ίδια μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν συμμορφώνεται με το πρότυπο έντυπο, το πιστοποιητικό γέννησης θα πρέπει να αναγνωρίζεται από άλλα κράτη-μέλη. Από τη στιγμή που ο πολίτης κατάφερε να εντοπίσει που βρίσκεται το έγγραφο, το μεταβιβάσει, το αναγνωρίσει επίσημα, το αναγνωρίσουν επίσημα, επόμενο εμπόδιο είναι το περιεχόμενο του εγγράφου οικογενειακής κατάστασης να αναγνωριστεί να μην έχει μόνο αναγνώριση του πιστοποιητικού γέννηση, να θεωρηθεί πιστοποιητικό γέννηση, αλλά να αναγνωρίζεται και το περιεχόμενο που αναφέρει το πιστοποιητικό γέννηση. Εδώ υπάρχουν τέτοια προβλήματα με τη μετάφραση και την επισημείωση, όπω ανέφερα, που μπορούν να εφαρμόζονται. Άρα μπορούμε να κάνουμε τι ίδιε συστάσει. Τα προβλήματα τώρα όσον αφορά την αναγνώριση του περιεχομένου ενό εγγράφου οικογενειακή κατάσταση. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει λόγω διαφορών όσον αφορά το εμπράγματο δίκαιο. Παραδείγματο χάρη, ε, τα διάφορα που αναφέρονται, τα στοιχεία που αναφέρονται στο πιστοποιητικό γέννηση ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οι γαλλικέ αρχέ μπορεί να αρνηθούν να αναγνωρίσουν ένα ιταλικό πιστοποιητικό γέννηση διότι δεν περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευκολύνει τη ζωή του πολίτη. Μπορεί να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν διάφορες ε, εξουσιοδοτήσεις να δέχεται βεβαιώσει ή να μπορούν ε, να αναγνωρίζονται τα έγγραφα παρά κάποιε ελλείψει που έχουν. Σύμφωνα, ε, υπάρχουν ελλείψει σύμφωνα με τον νόμο του χρο... της χώρας αποδοχής. Ε, άλλα προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν το περιεχόμενο του εγγράφου οικογενειακής καταστάσης μπορεί να σχετίζεται με τις διαφορές μεταξύ εμπραγμάτου δικαίου. Ας πούμε ένας ομοφιλόφιλος γάμος ολλανδικός δεν αναγνωρίζεται στην Ιταλία γιατί θεωρείται ότι είναι αντίθετος με την δημόσια πολιτική που ακολουθείται η γαλλική αναγνωρισμένη συμβίωση δεν αναγνωρίζεται στην Βουλγαρία διότι δεν ξέρουν ποιο είναι το νομικό οικοδόμημα που αναγνωρίζει αυτή τη συμβίωση. Όπως ακούσαμε από την προλαλήσασα, η αρμοδιότητα όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο είναι περιορισμένη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ίσως περαιτέρω δυνατότητα προσυζήτηση θα μπορούσε να εξή να δούμε τι δυνατότητες προσφέρονται από το άρθρο 21 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, αν η δράση την Ένωση είναι απαραίτητη και δεν, δεν παρέχει τι αναγκαίε εξουσίε ε, η συνθήκη, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω τη αναγκαία δικαιοδοσία που θα θεσπίσουν κανόνε για να διευκολύνουν την άσκηση τη ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό το άρθρο θα μπορούσε επίση να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένω και για το τελευταίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Ευρωπαίοι πολίτες, δηλαδή την αναγνώριση όχι μόνο του περιεχομένου συγκεκριμένου εγγράφου οικογενειακής καταστώσεως, αλλά και των συνεπειών που έχει αυτό το έγγραφο. Ας φανταστούμε ότι δύο Ιταλοί άντρε πήγαν στην Ολλανδία, παντρεύτηκαν και όταν επιστρέφουν στην Ιταλία και αξιώνουν κάποια ε, φορολογική ελάφρυνση που απορρέει από το ότι είναι παντρεμένο ζευγάρι, αυτό δεν εγκρίνεται διότι δεν αναγνωρίζεται ο γάμος τους που είναι γάμος ομοφιλοφίλων. Πέρα από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αλλάξει ε, η νοοτροπία όσον αφορά τα ομοφιλόφιλα άτομα και άτομα με διαφορετικούς ε, σεξουαλικούς προσανατολισμούς, ε, έχουμε δυνατότητες που προσφέρονται από το άρθρο 21 της Συνθήκης για της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ, δόκτωρα Έλλη Αντώνιο για την πολύ αναλυτική παρουσίαση αυτή που είναι τόσο ενδιαφέρουσα της μελέτης αυτής. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις ε, λύσεις που προτείνετε Καθώς και το ρόλο που προτείνεται για την Ένωση να ε, προσπαθήσει να ευνοήσει το διάλογο για το θέμα αυτό, αλλά να προωθήσει και λύσεις ε, βάσει το πρόγραμμα της Στοχόλμης για την δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Επόμενος είναι ο κύριος Duncan McNiven, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Προσωπική Κατάσταση. Είναι πρώην Γενικός Ληξίαρχος της Σκοτίας και θα μας μιλήσει για θέματα απάτης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Χαίρομαι που ε, είμαι εδώ, παρότι είναι έξι παρατέταρτο στο τέλος μιας μακριάς μέρας. Είμαι πρόεδρος λοιπόν αυτής της Διεθνούς Επιτροπής για θέματα οικογενειακής κατάστασης και όχι ως εκπρόσωπος του ε, Ηνωμένου Βασιλείου, γιατί όπω ξέρετε σήμερα είπε πολύ διαφορετικά πράγματα ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαι εδώ ω πρόεδρος αυτή τη Διεθνού Επιτροπή. Η οργάνωσή μας είναι λίγο γυρότερη από εμένα. Γεννήθηκε το 1939 με στόχο να ενθαρρύνει τη συνεργασία, με τη διεθνή συνεργασία και την ε, ανταλλαγή προφοριών για τα θέματα οικογενικής κατάσταση Έχουμε 15 χώρε μέλη, χώρε μέλη της Ένωσης και χώρε μέλη που δεν ανήκουν στην Ένωση. Και υπάρχουν μια σειρά από συμβάσει. Ορισμένε τις ανέφερε η δόκτωρ Έλλη Αντώνιο που μας ενδιαφέρουν. Επειδή μας ενδιαφέρει σε βάθος η ακρίβεια των ε, εγγράφων οικογενειακή κατάσταση μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα της απάτη. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας εδώ και χρόνια προσπαθεί να προλάβει φαινόμενα απάτη. Αλλά πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των ε, δράσεων για αποφυγή απάτης που πολλές φορές σημαίνουν περισσότερη αυτοκρατία, ελέγχους, ε, κοστίζουν, παίρνουν χρόνο και να διακρίνω λοιπόν μεταξύ αυτού και του κύριου καθήκοντός μας που είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης διακίνησης σε αυτές τις διαμεθεωρικές καταστάσεις που περιέγραψε η δόκτωρ Έλλη Αντώνιο. Αυτό είναι ο στόχος μας και δεν θέλουμε να υπάρχει ένταση μεταξύ αυτών των δύο στόχων, του κύριου και του δευτερεύοντος. Τι είδους απάτη υπάρχει στον τομέα αυτό δεν έχουμε πολλές ε, ακριβείς στατιστικές. Για παράδειγμα, πόσοι ε, παράνομοι μετανάστες, λάθρο μετανάστες υπάρχουν στο Βέλγιο. Δύσκολη απάντηση. Αλλά αυξάνει η απάτη αυτή όσο αυξάνει η διεθνής κινητικότητα. Και αλλάζει και η φύση της απάτης στον τομέα αυτό. Οι ληξίαρχοι σπάνια ε, κάνουν απάτες. Θα αναφέρω έναν δήμαρχο από μια χώρα που δεν την αναφέρω, που εξέδωσε ένα δικό του πιστοποιητικό θανάτου για να αποφύγει ποινική διαδικασία. Κυρίως ε, έχουμε φαινόμενα απάτης ε, όπως ε, ψευδείς δηλώσεις για λευκούς γάμους, ψευδείς αναγνωρίσεις πατρότητας. Κοιτάξτε, εμένα μου φτάνουν τα δύο παιδιά, αλλά ορισμένοι θέλουν πολλά παιδιά και αναγνωρίζουν ψευδός την πατρότητά τους και γενικώ ε, παραχαραγμένα ε, έγγραφα, κυρίως πιστοποιητικών γεννήσεως, ιδιαίτερα από κράτη εκτός ενώσεως, που δεν έχουν ε, αρκετά αξιόπιστα ληξιαρχικά αρχεία. Από το 92 η Ένωση προσπαθεί να προλάβει τέτοια φαινόμενα και το ίδιο και η οργάνωσή μας και χρησιμοποιούμε μια σειρά από όργανα. Έχουμε ακριβώς ε, τους ληξίαρχους ε, επιτόπου που ε, καταχωρίζουν τα στοιχεία και έχουμε και ειδικού επί του αστικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου από διάφορα πανεπιστήμια, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω. Έχουμε μία μόνιμη ομάδα εργασία για θέματα απάτη. Τελευταία συνεδρία έγινε τον ε, περασμένο Σεπτέμβριο, που συναντάτε που ε, συνεδριάζει ε, δύο φορέ το χρόνο και θα είναι το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς μας Γενικής Συνέλευσης τον προσεχή Μάρτιο. Συλλέγουμε πληροφόρηση με αυτά τα μέσα για τα είδη απάτης και τα αντίμετρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στον ένα τον άλλο βαθμό έχουν επιτύχει στα διάφορα κράτη-μέλη. Η, συστάση, η σύστασή μας 9 του 2005 χρειάζεται να αναφερθεί ως ιδιαίτερα σημαντική γιατί ταυτοποιεί τα χαρακτηριστικά των γνησίων εγγράφων και τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται η παρχάραξή τους. Συγκεκριμένα δηλαδή πρακτικά θέματα δεν έχουμε ωστόσο καμία πανάκια για να προλάβουμε την ε, απάτη και οι δράσεις που αναλαμβάνουμε έχουν περιορισμένα αποτελέσματα γιατί φυσικά δεν θέλουμε να θίξουμε τα ε, δικαιώματα των ανθρώπων σε προσωπική και οικογενειακή ζωή. Χρειάστηκε ε, να σεβαστούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να μην θίγουμε αυτά τα δικαιώματα. Είναι λοιπόν ανεπαρκής η προληπτική δράση. Τα αντίμετρα, τόσο προληπτικά όσο και τα... οι κυρώσει εκ των υστέρων, προωθούνται από τα κράτη, αλλά δεν μπορώ βέβαια να ισχυριστώ ότι είναι τέλεια αυτά τα μέτρα. Ποια είναι τα θέματα που απασχολούν την εργασία μας αυτή τη στιγμή. Την εργασία μας. Δύο θέματα. Το πρώτο προφανώς είναι η προσπάθεια να αποτρέψουμε την παραχάραξη εγγράφων ταυτότητας. Ελέγχοντας την ισχύ των ξένων εγγράφων ταυτότητας. Αλλά ιδιαίτερα ως άλλο κέντρο βάρου τη εργασία μας είναι η εργασία για να δημιουργήσουμε συστήματα πληροφορική που να μπορεί να ε, λειτουργήσει όπως ε, περιέγραψε προηγουμένως η δόκτωρα Ελιαντώνη. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε την ε, προσπάθεια πρόληψης της απάτης με την προσπάθεια ενίσχυσης της ελεύθερης διακίνησης. Διότι εάν μπορέσετε να παρουσιάσετε σε ένα ληξίαρχο ένα έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή, έγγραφο ταυτότητας, που βεβαίως είναι πολύ πιο δύσκολο να παραχαραχθεί. Αυτό το έγγραφο είναι πολύ πιο έγκυρο ενώπιον οποιοδήποτε ληξιάρχου από οποιοδήποτε άλλο πολύ απλούστερο έγγραφο που είναι πολύ πιο εύκολο να παραχαραχθεί. Τα ηλεκτρονικά συστήματα βοηθούν λοιπόν ε, την αντιμετώπιση της απάτης αλλά και την πρόληψή της, αλλά παράλληλα ευνοούν την ελεύθερη διακίνηση. Να κάνω τώρα και λίγη διαφήμιση για τη δουλειά μας, την περαιτέρω διαφήμιση, γιατί και η δόκτωρ Ελια Αντώνιο, την οποία δεν έχω συναντήσει προηγουμένως ε, και δεν τη δωροδόξα για να τα πει αυτά που είπε, αλλά ήταν πολύ καλή απέναντί μας, πολύ θετική. Έχουμε λοιπόν ε, τεράστια πείρα και ευρία έμπειρο γνωμοσύνη για θέματα οικογενειακής κατάστασης και όταν η Ένωση εξέδωσε τον Δεκέμβριο πριν από δύο χρόνια την πράσινη βίβλο για τα θέματα οικογενειακής κατάστασης. Ε, χάρηκα πολύ που είδα τα θετικά λόγια της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βεβαίως, εάν υπάρξουν νέες μορφές απάτης και αντιμετώπισης της, με χαρά συμμεριζόμαστε οποιαδήποτε εμπειρία. Βέβαια τα αντίμετρα αλλάζουν όπως αλλάζει και το είδος της απάτης. Τα μέτρα λοιπόν ε, που αναφέρονται στο έγγραφο που σας διένυμα συνεχώς αλλάζουν, ορισμένα μπορεί να μην είναι πλέον ε, χρήσιμα. Είπα λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικά συστήματα μηχανοργάνωσης και εκπώνησης ηλεκτρονικών εγγράφων. Πρέπει να το τονίσω ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο τμήμα, όχι όλο, το πρακτικό πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει και την ελεύθερη διακίνηση και να αντιμετωπίσει τις απάτες. Αυτό που χρειάζεται, κυρία Γερουσιαστή, είναι η πολιτική βούληση για να υπερβούμε κάποιες δυσχέρειες που ανέφερε και η δόκτωρ Ελή Αντώνιο τόσο αναλυτικά, ούτως ώστε να γίνει πιο ρωμαλαία η προσπάθεια των ληξιαρχείων και των κυβερνήσεων σε ολόκληρη την Ένωση για να προλαμβάνετε και να τιμωρείτε η απάτη στα έγγραφα οικογενειακής κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Μα καθόλου, μα καθόλου κύριε Μακλίβεν. Ήταν συναρπαστική η παρουσίασή σας. Και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο και στην αρχή και στο τέλος της παρουσίασής σας μας υπενθυμίσατε ότι όταν συζητάμε τα θέματα απάτη στον τομέα αυτό, ως ληξίαρχος και η οργάνωσή σας προσπαθείτε να ε, αντιμετωπίσετε από κοινού τα δύο πράγματα να συνδυάσετε την αντιμετώπιση της απάθης με την ελεύθερη διακίνηση. Αυτό είναι ζωτική σημασία, ε, να το σημειώσουμε όλοι. Και επίσης το άλλο που αναφέρατε. Τόσο φυσικά συνδυάσατε αυτά που είπατε με αυτά που είπε η κυρία Έλλη Αντώνιο. Επίσης το θετικό τρόπο με τον οποίο να τα θέματα αυτό, αυτά. Ότι μια ε, πλατφόρμα πληροφορικής που αναπτύσσεται μπορεί να βοηθήσει με θετικό τρόπο, ούτω ώστε ίσως ήδη να χρησιμοποιείται μάλιστα, όπως είπατε, για να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Και επίσης αυτή η έκκληση που κάνετε για πολιτική βούληση, πολύ σωστό, σχεδόν τα έχουμε καταφέρει. Θα μπορούσαμε να ε, καταλήξουμε αλλά ε, διορθώνει, συμπληρώνει ο κύριος Μακνίβεν, αυτή η πλατφόρμα είναι στο τελικό τη στάδιο. Συγχρηματοδοτήθηκε μάλιστα από την Ένωση. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ζαπών. Θα υπάρχουν ερωτήσεις, ε, είμαι σίγουρη. Αλλά ας περάσουμε στον τελευταίο μιλητή μας, την δόκτορα Μπογιάννα Ζάντραβεκ, που θα μιλήσει για τα έγγραφα προσωπικής κατάστασης, οικογενειακής κατάστασης, πώς θα μπορέσουν να υπερβούν τα ληξιαρχεία τα προβλήματα που προκύπτουν από νομοθετικά κενά. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τα προβλήματα των ληξιάρχων ε, και την προσπάθεια υπέρβασης των προβλημάτων που οφείλονται σε νομοθετικά κενά. Ε, κατάγομαι από το Μάριμπορ, τη δεύτερη πόλη της ε, Σλοβενίας και εργάζομαι ως λεξιάρχος εδώ και 25 χρόνια. Ε, είμαι αρκετά εξοικειωμένη, έως πολύ εξοικειωμένη με τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνώνυμο τη σύγχρονη κοινωνία. Όχι όμω, δυστυχώ, στον τομέα τη οικογενειακή ή προσωπική κατάσταση. Οι διαφορέ στι νομοθεσίε για την προσωπική κατάσταση μεταξύ των χωρών μελών είναι πολύ μεγαλύτερε τώρα από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Οι Ευρωπαίοι πολίτε ε, αντιμετωπίζουν πολλέ διοικητικέ δυσκολίε όταν προσπαθούν να δηλώσουν την οικογενειακή του κατάσταση. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνε ε, σε σχέση με τις προσωπικές καταστάσεις και αυτό οδηγεί σε ε, διάκριση και παρεμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους στα πλαίσια των κρατών μελών διαφορετικές νομοθεσίες και διαφορετικός τρόπος πρόβλεψης και μεταβολής της προσωπικής κατάστασης, διαφορετικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ή την διακοπή διαφόρων σχέσεων, διαφορετικοί τρόποι καταγραφής της προσωπικής κατάστασης και τα διαφορετικά έγγραφα είναι μερικά μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες και με τα οποία πρέπει να ζήσουν. Για παράδειγμα, ένα ε, παιδί που έχει διαφορετικά επώνυμα σε δύο χώρες μέλη. Ε, έχουμε έγγραφα ε, για το ίδιο παιδί που αναφέρουν διαφορετικούς γονείς σε κάθε κράτος μέλος, γιατί έχει δηλωθεί το ονοματεπώνυμό του σε ένα... και έχει μεταβάλει το ονοματεπώνυμό του σε μια χώρα, αλλά δεν μπορεί να, μεταφέρει... να μεταφέρει αυτή τη μεταβολή σε άλλη χώρα μέλος. Επίσης, ε, σε ομοφυλόφιλα ζευγάρια ή σε καταχωρημένες ε, σχέσεις συμβίωσης. Ε, σε χώρες που δεν αναγνωρίζεται σχέση συμβίωσης, κάποιος που είναι παντρεμένος σε μια χώρα αναγνωρίζεται ως άγαμος, ως μη, μη δεσμευμένος άλλη χώρα. Και επίσης υπάρχουν διαφορετικά έγγραφα στα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, Υπάρχουν έγγραφα που δεν εκδίδονται καν από μερικές χώρες μέλη. Και μάλιστα χώρες που δεν έχουν συνάψει αμοιβέ συμφωνίες ε, για την αμοιμοποίηση, αυτό με την νομιμοποίηση των εγγράφων, απαιτούν ε, αποσπάσματα ή ληξιαρχικές πράξεις ε, με, με γενικά έντυπα και μερικές φορές απαιτούν και συμβολιογραφικά έγγραφα. Και μάλιστα και η μεταβολή του, της προσωπικής κατάστασης μερικές φορές πρέπει να περνά από διπλωματικές διάβλους που είναι πολύ χρονοβόρες. Όταν δεν έχουν ε, συναυθεί διμερείς αμοιβές συμφωνίες για την ανταλλαγή δεδομένων, ε, τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να κοινοποιούν τις μεταβολές της οικογενειακής κατάστασης ε, των πολιτών που λαμβάνουν χώρα στο δικό τους έδαφος. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και τα κοινωτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να προσπαθήσουν να άρουν τα προβλήματα που δημιουργεί αναγνώριση της προσωπικής κατάστασης του ατόμου. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ενοποίηση ε, στα θέματα προσωπικής κατάστασης ε, στα κράτη-μέλη έχει επίγοντα χαρακτήρα και η διαδικασία ενοποίησης των εθνικών νομοθεσιών ε, θα ήταν επίσης ευπρόσδεκτη. Μια όμως και υπάρχουν προβλήματα στα θέματα μεταβολής και καταγραφής της οικογενειακής κατάστασης είναι τα πιο σημαντικά τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, αν θέλουν να επιλύσουν έστω και εν μέρη τα προβλήματα αυτά, θα πρέπει να δράσουν κατεπηγόντως, να ε, θεσπίσουν κάποια μέτρα, τουλάχιστον ε, να μετρι... για να μετριάσουν την παρούσα κατάσταση. Μερικά από αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ήταν τα εξή. Τα μέτρα αυτά ταξινομούνται ανάλογα με την δυνατότητα εφαρμογής τους. Εξάλληψη της ανάγκης για έκδοση εγγράφων συμβολογραφικού τύπου στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το λόγο μέτρο απλώς με την επίτευξη αμοιβαία συμφωνίας. Άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τυχόν μεταβολές στην προσωπική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, τις οποίες η χώρα στην οποία το άτομο άλλαξε την προσωπική του κατάσταση θα πρέπει να υποβάλει στη χώρα στην οποία το άτομο γεννήθηκε και της οποία έχει την ηθαγένεια. Και αυτό το μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σχετικά γρήγορα Απαιτείται απλώ μια συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων που τηρούν το αρχείο της προσωπικής κατάστασης ενός ατόμου στα επιμέρους κράτη-μέλη. Θέσπιση ενός ενιαίου εντύπου για την καταχώρηση των μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση. Μία εναλλακτική λύση θα ήταν η εισαγωγή ενός εντύπου που θα περιλαμβάνει ε, τα δεδομένα αυτά στα, στη γλώσσα της χώρας που εξέδωσε το έγγραφο και στα αγγλικά ταυτόχρονα. Αναγνώριση των ονομάτων, όνομα και επώνυμο που οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν σε άλλο κράτος μέλος. Εναρμόνιση των αλφαβητικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται κατά την καταχώρηση της προσωπικής κατάστασης και για το μέλλον ίσως δημιουργία ενός ε, Μητρώου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσωπική κατάσταση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα τροφοδοτούν τα κράτη-μέλη με τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση και αναγνώριση της προσωπικής κατάστασης που ένα άτομο έχει αποκτήσει ή απολαμβάνει σε ένα κράτος μέλος από όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια για τη ρύθμιση του θέματος της οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των νομοθετικών κενών που παρατηρούνται στον ελόγο τομέα. Μία λύση θα ήταν η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη ρύθμιση του ελόγω τομέα από τα κράτη-μέλη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο των χωρών που ρυθμίζουν το θέμα της οικογένειακή κατάσταση με φιλελεύθερο και ανοιχτό πνεύμα, καθώς και να καταγράψει τις αλλαγές στον τρόπο ζωής και στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Ως ληξίαρχος λοιπόν είμαι υπέρ των ε, δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέτρων προκειμένου να ρυθμιστεί το θέμα της προσωπικής κατάστασης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ήδη επισήμανε την ε, μεγάλη σημασία μιας ε, ενιαίας κατάστασης, προσωπικής κατάστασης, ενιαίου συστήματος προσωπικής κατάστασης και επίση η, αναγνώριση των νομίμως κατοχυρωμένων εγγράφων πολιτικών οικογενειακής κατάστασης ε, είναι σημαντική για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Εμείς ε, στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στον τομέα αυτό και είμαστε πρόθυμοι για συνεργασία και συνδρομή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν της πολυπόθητης ενοποίησης της ρύθμισης για την προσωπική κατάσταση, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη της αμοιβαίας αναγνώρισης, αυτόματης αναγνώρισης των νομίμων εγγράφων, χωρίς ανάγκη συμβολιογραφικών επιπλέον εγγράφων και μεταφράσεων. Και επίσης ε, άμεση ανταλλαγή των ληξιαρχικών πράξεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Και μόνο με αυτέ τι λύσει θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε τι διαδικασίε για την καταχώρηση μεταβολών οικογένειακή κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών. Και με ιδιαίτερη χαρά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ληξιάρχων θα παράσχει πληροφορίες για διαδικασίες σε θέματα προσωπικής κατάστασης ε, αν χρησιμοποιηθούν αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλύσει τα προβλήματα που επισημάναμε στο εγγραφό μας. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ, Δόκτωρα Ζάντοβεκ. Έξοχη παρουσίαση ακόμα μία και συμπληρώνεται άριστα τους προηγούμενους συναδέλφους στις πρώτερες παρεμβάσεις τους και σωστά τονίσατε το θέμα της ενοποίησης, της κοινή αντιμετώπισης όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση και το... αυτό ε, χτύψε κάποια χορδή μέσα μου. Αυτό σημαίνει τι, μπορεί, τι σημαίνει να είναι κανείς κράτος μέλος, μέλος. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, περισσότερο κοινό έδαφος που καλύπτει ε, τους πολίτες μας σαν μέλη κοινότητας, σαν μέλη οικογένειας. Ε, δόθηκαν, προτάθηκαν πολλές λύσεις τα προβλήματα, πιστεύω, από αυτά που υπόθηκαν. Και πιστεύω ότι με τα χαρά θα άκουγα κάποια σχόλια ή τυχόν ερωτήσεις που έχετε. Ε, όμως, αν εντοπίσετε και άλλα προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν και λύσεις. Θα δώσω το λόγο σε εσά τώρα. Παρακαλώ να συστηθείτε καταρχάς και μετά να υποβάλλετε τυχόν ερώτηση, σχόλιο. I understand is that of the European Commission. Κάποιος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλετε κάτι, ίσως κάποια συνεισφορά κάποιον στη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σάλα μου είναι με λένε. Είμαι επικεφαλής της μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης στο θέμα του πολιτικού, του αστικού δικαίου. Ευχαριστώ τους πολίτες και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Ακούσαμε πολλές ιδέες, ακούσαμε και διάφορες λύσεις που προτάθηκαν και ευχαριστώ τους ομιλητές γι' αυτό. Τώρα στο τελευταίο τμήμα αναφέρθηκαν ζητήματα πολύ γνωστά. Από το 2007 τα μελετούμε και έχουμε ετοιμάσει παρόμοιες μελέτες με αυτές που ετοιμάζεται τώρα για την οικογενειακή κατάσταση το επόμενο, υπάρχει γνώση. Επόμενο βήμα. Πώς τεχνικά και πολιτικά θα είναι εφικτό να βρούμε λύσεις. Και στο παρόν νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θεσπίζεται τις συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί της βάσεως του προγράμματος της Στοχόλμης και του σχεδίου δράσεως της Στοχόλμης. Συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία νομοθετικών πρωτοβουλειών που αφορά την μεταβίβαση δημοσίων εγγράφων για διοικητικές ε, διαδικασίες. Κάτι που αφορά αυτά που έθιξε η κυρία Ηλιαντώνιο και δεύτερον, δεύτερη πρωτοβουλία προβλέπουμε για τις συνέπειες της αναγνώρισης εγγράφων οικογενειακής κατάστασης. Έγινε δημόσια διαβούλευση το 2010 και το 2011 για αυτά τα ζητήματα. Συνεχίζεται η προσπάθεια και οι εργασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, τι ήθελα να πω κάτι, συγκάτσα κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Η πολιτική πτυχή. Ναι, πράγματι πρέπει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στο επίπεδο των πιο φιλελευθέρων κρατών μελών. Αυτό αναφέρθηκε. Πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε Ένωση 27 κρατών μελών και όλα τα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει το επίπεδο της προσφοράς τους προς τους πολίτες. Στόχος της Ένωσης είναι να βρει κάτι επί το οποίο μπορούν να συμφωνήσουν οι 27 ή τουλάχιστον επαρκής πλειοψηφία των 27 κρατών μελών βάση των κανόνων της συνθήκης. Άρα, κατά την άποψή μου, πρέπει να βρούμε τον κοινό παρανομαστή που μπορεί να προσφέρει τη λύση. Αυτό θα διευκόλυνε την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, κάτι που συζητήσαμε σήμερα. Προσπαθήσαμε στις δημόσια βουλεύσεις να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Πολλοί παριστάμενοι στην αίθουσα τροφοδότησαν τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Νομική Επιτροπή που επίσης δίνει τροφή προσκέψη και τροφοδοτεί τις εργασίες που κάνουμε για ένα θέμα που είναι τόσο επίκαιρο όπως αυτή η οικογενειακή κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, για τα σχόλιά σας και άλλοι θα θέλουν να σχολιάσουν αυτά που είπατε. Επόμενος, ορίστε, έχετε το λόγο. Εγώ προτιμώ να κάνω μία μικρή πρόταση όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πράξεων στα κράτη-μέλη. χρησιμοποιώ τη δική μου εμπειρία. Εργάστηκα σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Χρειαζόμουν διάφορα τέτοια έγγραφα και πιστοποιητικά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είμαι Γερμανή υπήκο. Κατοικώ στην Ολλανδία. Και χρειάζομαι την, ε, το πιστοποιητικό γέννηση όταν πάω στη Γερμανία για να πάρω το πιστοποιητικό γέννηση μου δίνει ταυτόχρονα και μια μετάφραση σε μία από τις τρεις γλώσσες που είναι οι πλέον ομιλούμενε στην Ευρώπη. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, φερρυπίν. Είναι ένα παράδειγμα και μόνο αυτό. Και αυτή η μετάφραση γίνεται, είναι γραπτή και είναι απαραίτητη για να την παρουσιάσω, να την υποβάλω στην Ολλανδία. Πληρώνω ένα φόρο για αυτή τη μετάφραση στο φορέα τον αρμόδιο. Είναι αναγνωρισμένη νόμιμη αναγνώριση, κρατικός φορέας γερμανικός κάνει τη μετάφραση, χρειάζομαι λιγότερο χρόνο γιατί υπάρχει ήδη μετάφραση, μπορώ να πάρω το έγγραφό μου και να πάω με αυτό το πιστοποιητικό και να το παραδώσω στις αρμόδιες αρχές της Ολλανδίας. Αυτό είχα να πω, αυτό είναι το σχολείο μου. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Υπάρχει κάποιος που θέλει να υποβάλει κάποιο σχόλιο, να ρωτήσει κάτι. Ορίστε, εκεί πίσω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω γαλλικά. Είχα μία ερώτηση να κάνω. Αναφέρθηκε αυτό που θέλω να θίξω. Για να προχωρήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεω. όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ανάγκη να βρούμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν συνεπάγεται το να ανακαλύψουμε τη συνέπειες ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και θέτω το ερώτημα. Εκεί που βρισκόμαστε τώρα, εκεί που φτάσαμε και θέλουμε να κατασκευάσουμε μια πολιτική ένωση που πλησιάζει τον πολίτη. Μήπως πρέπει να ξεπεράσουμε και αυτά που αποτελούσαν την καρδιά των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να ξεπεράσουμε το όραμα που αφορούσε, επικεντρωνόταν στην ελεύθερη μετακίνηση και να πάμε σε κάτι που πηγαίνει πιο μακριά. Ένα πολιτικό πρόγραμμα, οικοδόμημα. Ποια είναι η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε. Προτείνοντας το εξή κατά την απόψή μου. Η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι της διαφοράς, της πολιτισμικής διαφοράς, της ποικιλία όσον αφορά τα οικογενειακά θέματα. Και αν το νέο αυτό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην αφορά ένωση και ομοιομορφία αποκλειστικά της μετακίνησης. Αντιθέτως, να βρούμε έναν τρόπο να συντονίσουμε τη διαφορά που υπάρχει, τις διαφορές που υπάρχουν για να τις διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα οικοδόμημα πολιτικό που θα εδράζεται επί της ποικιλομορφία. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Θα επιστρέψω στα μέλη του πάνελ τώρα και θα σας παρακαλούσα να σχολιάσετε τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν και αν έχετε να πείτε κάτι τελικό, έτσι θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που υπόθηκε, το ερώτημα που υπευλήθη. Ίσως έχω φιλοσοφική προσέγγιση των πραγμάτων, θέτεται θέμα πολιτικής φιλοσοφίας, ίσως αυτό πρέπει να εξεταστεί επίσης, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε εκεί ή και με την πρακτική καθημερινή ζωή. Από οποιαδήποτε πλευρά καταλήγουμε στο ίδιο σημείο τελικά. Λύσεις, βελτιώσεις. Ξεκινάμε λοιπόν από τον κύριο Μακνίβεν. Ευχαριστώ πολύ. Να αντιδράσω στους τρεις που πήραν το λόγο από την Επιτροπή με την οποία συνεργαζόμαστε πολύ στενά θα ενεθάρρυνα την Κομισιόν στην εργασία της που νομίζω ότι θα καταλήξει να επιτύχει. Πέπρωτε να επιτύχει τους στόχους που ανέφερε η κυρία Ελιαντώνιο. Νομίζω ότι η Σέλα και οι συνάδελφοί της διαπίστωσαν ότι ήταν περίπλοκη η κατάσταση. για το πώς να αντιμετωπίσουμε τα πρακτικά προβλήματα ξέρουμε, αλλά την πολιτική κατάσταση είναι πιο δύσκολο. Θέλει χρόνο. Καλό λοιπόν την Κομισιόν να συνεχίσει, να εμείνει γιατί αξίζει τον κόπο. Και φυσικά μπορεί να βασιστεί στη βοήθεια της Ένωσης των Ληξιάρχων, όπως είπε η συνάδελφός μου, στην δική μου επιτροπή και πολλούς άλλους ειδήμονες ο κύριος από το Παρίσι σωστά περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Την δυσχέρεια που αντιμετωπίζουμε. Τι είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Φιλοσοφικό θέμα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου το έθιξε νωρίτερα σήμερα. Δεν θα ήθελα να μπω στα χωράφια του. Μιλήσατε για πολιτιστική πολυμορφία επίσης. Αυτή η πολιτιστική πολυμορφία που εγώ ως Σκοτσέζος από την άνω αριστερά αγωνία της Ευρώπης θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν εμποδίζει τους ε, πολιτικούς μας στην προσπάθειά τους επίτευξης κοινή οδού πρόοδου. Οι Γάλλοι για λόγους πολιτιστικούς ε, απόλυτα κατανοητούς αγαπούν ε, τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τα θέματα των ε, ονομάτων και επωνύμων. Αυτή λοιπόν η πολιτιστική πολυμορφία αντιτίθεται κάπως στα πιο ομοιογενή συστήματα που οι τρεις ειδήμονες εδώ προτείνουν. Για την Γερμανίδα κυρία που ζει στο Βέλγιο και δεν θυμάμαι σε ποια τρίτη ε, χώρα αναφέρθηκε. Πολύ καλό παράδειγμα της ε, συγκεκριμένης πρόοδου που έχει επιτευχθεί από τις εθνικές αρχές και όπως είπε και η δόκτωρα Ηλιαντώνιο η αρχή η δική μας έχει μία πολυγλωσσική αντιμετώπιση παρέχει δηλαδή τα πιστοποιητικά της σε διάφορες γλώσσες. Έχουμε μια σύμβαση που έχουν υπογράψει 20 χώρες, κάποια κράτη-μέλη και κάποια μη-μέλη έχουν υπογράψει, αλλά είναι μόνο 20 χώρες. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους. Και τα ωφέλη που ε, διεπίστωσε η Γερμανίδα συναδελφός μας θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε άλλους. Δεν ξέρω τι θέλουν να, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ έξοχα. Σίγουρα μπορεί να θέλουν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να πω μόνο ότι ξέρω ότι οι ιδέες μου είναι λίγο ευρύτερες από το τωρινό πλαίσιο, αλλά ξέρω ότι πολλοί δεν μένουν ε, στη χώρα της οποίας έχουν την ηθαγένεια. Γιατί να μην τους επιτρέψουμε να ζουν όπως ακριβώς επιθυμούν. Γιατί κλείνονται οι χώρες πίσω, οχυρώνονται πίσω από τις παραδόσεις τους για θέματα οικογενειακού δικαίου, σχέσεων ε, μεταξύ δύο ατόμων. Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι παραδόσεις. Γιατί δεν εμπιστεύονται κάπως περισσότερο τα, τους ανθρώπους μέσω πιο φιλελεύθερων νόμων για να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι όπως θέλουν. Για να μην χάνουν εξουσία τα κράτη. Κάτι πρέπει να κάνει η Ένωση. Γιατί υπάρχουν όντως προβλήματα και κάποια προβλήματα εύκολα, πραγματικά εύκολα θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, να επιληθούν. Ευχαριστώ. Μα ολόψυχα συμφωνώ. Οι παραδόσεις πρέπει να είναι κάτι το ζωντανό αλλά σε επανέλθουμε στην ε, δόκτορα Έλλη Αντώνιο. Τρεις παρατηρήσεις, καταληκτικές. Μα φυσικά συμφωνώ με τον κύριο Μακνίβεν. Τεχνικές λύσεις έχουμε. Αλλά το θέμα είναι η πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν. Δεύτερον, να αντιδράσω στους δύο προηγούμενους. Βεβαίως Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ ε, θεωρητικών αντιμετωπίσεων και πρακτικών προβλημάτων. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε τι είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η πολυμορφία κτλ. Αλλά στην πράξη αυτό που παίζει ρόλο για τον καθένα μας ως πολίτη της Ένωσης είναι πόσα ταξίδια πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως. Μπορούμε να παντρευτούμε. Μπορούμε να ε, έχουμε πρόσβαση σε κάποια επιδόματα. Βεβαίω, ο στόχο είναι να λύσουμε πρακτικά προβλήματα. Και τέλος, τέλος, η συζήτηση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα από τη μία και την εθνική ταυτότητα από την άλλη, αλλά αξία δεν είναι μόνο η ταυτότητα, αλλά και η αποδοχή των άλλων, η αποδοχή της ταυτότητας των άλλων. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε, αλλά να αναγνωρίζουμε την ταυτότητά του, να την αποδεχόμεθα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε ενδεχομένω τη συζήτηση. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Αλλά νομίζω ότι με χαρά όλοι θα συμφωνήσουν να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας.